Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Ζητώ συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση. Per favore, se volete sedere. Παρακαλώ να καθίσετε για να αρχίσουμε με τι εργασίε μας με την ηλεκτρονική ψηφοφορία της έκθεση Βόμποντα. Sulla ε, Passiamo allora. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Νομίζω ότι μάλλον έχει απορριφθεί. Θα ήθελα όμως να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε με την κάρτα σας. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ψήφισαν 30 υπέρ, 26 κατά. Δύο αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Ας προσπαθήσουμε. 14. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Λείπουν και μερικοί. Ισοψηφία. Άρα απορρίπτεται. 27 υπέρ, 27 κατά 15 παρακαλώ δεν έχω την κάρτα μου μαζί να με συνυπολογίσετε Θέλετε να ψηφίσετε για τη 13, ρωτάει ο πρόεδρος. Υπέρ. 28-27, άρα εγκρίνεται. Ψηφίζαμε τη 13, λέει ο πρόεδρος, με συγχωρείτε. Με την ψήφο του συναδέλφου έχουμε 28-27, άρα περνάει 14. Υπέρ. Μα την έχουμε ψηφίσει τη 14. Corretto έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Συμβιβασμός 1. Θέλετε να ελέγξουμε τη 16, αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 16. Υπάρχουν ε, πέντε που έχουν βάλει την κάρτα τους αλλά δεν ψηφίζουν. Α, τώρα είναι τέσσερις. Σε πάση περιπτώσει, αποφασίστε. Περίεργο. 32 υπέρ, 27 κατά. Δύο αποχές. Εγκρίνεται. Συμβάσμα 1. Πρώτο τμήμα. Τάνο. Πρόεδρε. Ο κύριος Βόμποτα συμφωνεί ως προς τη σύνταξη, γιατί όταν το διάβασα δεν ήταν σαφές όταν μιλούσαμε για ενδυνάμει, ενδυνάμει επιπτώσεις διαφθοράς θα μιλάμε για παρεπόμενη διαφθορά μέσα στα πλαίσια των θεσμικών οργάνων. Είναι θέμα συντακτικό καθαρά στα αγγλικά. Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, Εχθές ε, στις πολιτικές ε, ομάδες, οι πολιτικές ομάδες διαπραγματεύτηκαν για αυτή την συμβαστική πρόταση και είπαμε χθες με σαφήνεια στην Επιτροπή ότι είμαστε υπέρ των ε, συμβασμών εκτός από το δεύτερο τμήμα του 1 και του 6. Και από εχθές σε αυτή τη συμβαστική πρόταση 1 μυστικά προσθέθηκε μία πρόταση στο πρώτο τμήμα στο οποίο, στον κατάλογο της ψηφορία μας αυτό το πρώτο αναφέρεται ως δεύτερο και πρόκειται για τον ισχυρισμό του κυρίου Φέρν ότι ε, θα μπορούσε να υπάρχει διαφθορά και στους ε, θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια τόσο τεράστια καταγγελία που παρακαλώ τον κύριο Φέρν είτε να καταθέσει αποδείξεις για αυτό το θέμα, για τον ισχυρισμό του, είτε να ψηφίσει μαζί με εμά. Να συμφωνήσει με εμά. Γιατί, ξέρετε, βλέπω ότι θα δημιουργηθεί πολιτικό ζήτημα. Να προβλέπονται, να συμπεριλαμβάνονται καταγγελίε ε, τόσο σημαντικές σε ένα θέμα χωρίς να έχει υπάρξει διαπραγμάτευση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ε, διαμαρτύρομαι όσον αφορά τη διαδικασία. Μέχρι τώρα η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα συναδελφική, αλλά αυτό πλέον δεν ισχύει και παρακαλώ τους συναδέλφους να ψηφίσουν ε, μόνο το υπαρθμόν 1 και να καταψηφίσουν το σημείο 2 και το σημείο 3. Ο κύριος Βόμποντα. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η πρόταση βασίζεται σε μία τροπολογία που περιλαμβάνεται στι τροπολογίε, Αυτό δεν είναι και ναι αυτή η πρόταση. Όμως θέλω να προτείνω το εξή, κύριε Πρόεδρε. Αυτή την πρώτη παράγραφο να την ψηφίσουμε χωρίς αυτή την πρόταση και όσον αφορά αυτή την πρόταση να την ψηφίσουμε ξεχωριστά. Γιατί έχει δίκιο ο κύριο Πόσελ, δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχή ε, και γι' αυτό ε, ας ακολουθήσουμε ε, την τον κατάλογο ψήφου. Πράγματι, λέει ο Πρόεδρος, ας ψηφίσουμε για το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Με την προφορική μου όμως τροπολογία, εντάξει. Κατά αποχές. Υπέρ του πρώτου τμήματος λοιπόν. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα γιατί δεν είναι καθόλου σαφές. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Πέντε δεν ψήφισαν. 33 υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. 24 λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Θα ήθελα να ελέγξουμε η ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 25. Έξι δεν ψηφίζουν. 33 υπέρ, 29 κατά εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, μου φαίνεται ότι απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2. Ωραία, ελέγχουμε την 29. Τέσσερις δεν ψηφίζουν. Τι να κάνουμε. 35 υπέρ, 27 κατά, εν μία αποχή εγκρίνεται. δύο υπέρ του συμβασμού δύο κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβασμού 3. Άμε συγχωρείτε 32 υπέρ, κατά. Ψηφίσουμε την 32. 32. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά, αρχίζει η ψηφοφορία επί της 32. Ψηφίζουμε. Πέρας. 19 υπέρ, 44 κατά. Απορρίπτεται. Σαφώς. Τροπολογία συμβασμού 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία συμβασμού 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 6. Ονομαστική κλίση. Πέρας. 36 υπέρ, 30 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία συμβασμού 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ του συμβασμού 8 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά δεν είναι σαφές. Δεύτερο τμήμα, της 53 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Chiusa la votazione. Πέρας. Απορρίπτεται 49 κατά 15 υπέρ. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 14, τροπολογία 57 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 56. Ε, Ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία. 39 υπέρ, 28 κατά. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της 56 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Όχι. Ας ελέγξουμε λοιπόν. Τρίτο τμήμα. Αρχίζει η ψυχοφορία επί του τρίτου τμήματος της τροπολογίας 56. Πέρας. Πέντε κάρτες περισσότερες από τους ψηφίσαντες. 38 υπέρ, 28 κατά εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται 69 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία συμβιβασμού 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 73 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται νομίζω. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 73. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 38 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ της τροπολογίας συμβασμού κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 τροπολογία συμβασμού 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 83. Είναι προφορική. Όχι, λέει ο πρόεδρος. Με συγχωρείτε. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. 80... Θέλετε να ελέγξουμε. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ci sono 70 schede inserite. Έχουμε 70 κάρτες και έχουν ψηφίσει μόνο 60 συνάδελφοι. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία, αλλά 9 ε, συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Τώρα είναι 7. Δηλαδή έχετε εισαγάγει την κάρτα σας αλλά δεν έχετε ψηφίσει. Επτά από σας. Ωραία. Κλείνουμε την ψηφοφορία. 35 υπέρ, 28 κατά. Τροπολογία συμβιβασμού 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι σαφές. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ελέγχουμε για την 4. Ψηφίστε παρακαλώ. Τροπολογία 4. Πέρας, 31 υπέρ, 33 κατά, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά. Και εδώ δεν είναι σαφές, μάλλον απορρίπτεται, αλλά δεν, είμαστε, δεν είμαι σίγουρος. Απορρίπτεται. Εντάξει. Τώρα ψηφίζετε περισσότερο Ψηφίζουμε την 5, 5 ηλεκτρονικός έλεγχος. debito. Μερικοί δεν ψήφισαν. 49 κατά, 15 υπέρ. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την έκθεση. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Να bene. Τι έχει chiudi. Va bene, 62 favore. 62 υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές. Να συγχαρούμε τον εισηγητή, τον κύριο Σφόβοντα. Λοιπόν, Allora, qualche, qualche indicazione sull'ordine di voto. Να πούμε ορισμένε στοιχεία σχετικά με την ψηφοφορία για το επόμενο θέμα Καλούμεθα λοιπόν να ψηφίσουμε για, ένα, ε, για την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Συμφωνία Σύμπραξης ε, με το Τουρκμανιστάν και κατόπιν ε, θα ψηφίσουμε για την πρόταση ψηφίσματος. Μετά στο τέλος θα ψηφίσουμε για την πρόταση της κυρίας Άουταλα να συστήσουμε στήσουμε στην Ολομέλεια προς το παρόν να ανασταλεί η ψηφοφορία για την συμφωνία και να περιμένουμε να γίνει το ταξίδι στο Τουρκμενιστάν το Μάιο, να πάει η αντιπροσωπεία μας και μετά να ψηφίσουμε. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι εδώ πρόκειται μόνο για μία σύσταση, για μία αξιολόγηση πολιτική ε, κατά πόσον αυτά τα οποία ε, προτείνονται ε, στην Ολομέλεια αντιστοιχούν με τις επιθυμίες των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία για τη σύσταση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας. Όσον αφορά τις τέσσερις πρώτες τροπολογίες, αυτές είναι ταυτόσιμες, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται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 Πρέπει να περιμένουμε λίγο γιατί έχουμε 69 κάρτες που έχουν ε, εισαχθεί και έχουν ψηφίσει μόνο 61. Μα γιατί ψηφίζουμε, λέει ο κύριος Άτκινς, για ποιο πράγμα ψηφίζουμε, πρόεδρος. Ψηφίζουμε για τη σύσταση της ε, κυρίας Νικολάη. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας. Ε, Λείπουν 8. Λείπουν 7. Κλείνουμε όμως την ψηφοφορία. 51 υπέρ, 9 κατά, 2 αποχές, εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε για την πρόταση ψηφίσματος Ξεκινάμε με την τροπολογία υπερθμών 25. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται 27 όχι 24 λέει ο πρόεδρος εγκρίνεται ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 24 λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το 24. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 24, παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία για την 24. 35 υπέρ, 32 κατά. Εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 μαζί με την 34 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 33 ε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται δεν ψηφίζουμε για την 35 γιατί έχει ήδη καλυφθεί από την προφορική τροπολογία. 36 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 41. Μισό λεπτό, 37 λέει τώρα ο πρόεδρος. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 38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 αποχές εγκρίνεται. 45 και 46 είναι ταυτόσημες, ως εκ τούτου υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 47-48 ε, καταπίπτουν, πάμε στην 49, υπέρ παρακαλώ, κατά, δεν είναι σαφές, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά Ψηφίζουμε για την 49 ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λείπουν μόνο δύο ψήφοι, κλείνει η ψηφοφορία. 36 υπέρ, 26 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές απο... εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 81 υπέρ κατά εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά δεν είναι σαφές ηλεκτρονική ψηφοφορία ελέγχου για την τροπολογία 83 άρχεται η ψηφοφορία έκλεισε η ψηφοφορία 40 υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, ούτε και αυτό μου είναι σαφές. Αν δεν σηκώνετε τα χέρια, πώς να καταλάβω. Ξεκινάει λοιπόν η ψηφοφορία για την 85 το συγγνώμη που χάνουμε χρόνο, αλλά και εσείς αν δεν σηκώνετε το χέρι, εγώ που να ξέρω για ποιο τι, τι πράγμα ψηφίζετε. Λοιπόν, τρεις ε, συνάδελφοι ξεχνάνε να ψηφίσουν, έκλεισε η ψηφοφορία. Ε, αποτέλεσμα, 27 έως 40. Ε, Βλέπετε, εγκρίθηκε με ε, μεγάλη πλειοψηφία, άρα έπρεπε να έχει σηκώσει το χέρι. Επόμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 89, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 7 συμβαστική σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, θα έλεγα εγκρίνεται η 8 η συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η εννέα συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 129 τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Οι 130 και 131 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε και για τις δύο υπέρ, κατά, Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική ψηφορία ελέγχου για τις 130 και 131. Ψηφίζουμε. Συνεχίζουν τρεις, άντε δύο τώρα στην άλλη να μην ψηφίσουν. Έκλεισε η ψηφορία. Ε, το αποτέλεσμα 27-40 ε, είναι σαφή ε, συντριπτική η πλειοψηφία. Τι να πω. Η 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 133 υπέρ κατά αποχές ε, νομίζω απορρίπτεται. Όχι. Λοιπόν, έλεγχος για την 133. Ψηφίζουμε. 39 υπέρ, 28 ε, κατά, υπέρ κατά, για την 134 τώρα, εγκρίνεται, η 135 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω απορρίπτεται, η 136 Θέλετε έλεγχο? Όχι. Λοιπόν, 136. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 134 144 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι 153, 54 και 55 είναι ταυτόσιμες ε, υπέρ, ε, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Οι 156 υπέρ, κατά, απο αποχές απορρίπτεται. Η 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 158 159 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίπτεται αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Οι 159 ε, ψηφίζουμε. Chiusa la votazione. 39 a 28 è approvato. 160 voti favorevoli. 160 υπέρ. Contra. Κατά. Αποχές. Εγκρι... Ε, βλέπω λοιπόν ότι και εδώ ε, ψηφίζεται με τον ίδιο τρόπο, έστω και αν σηκώνεται τα χέρια διαφορετικά. Εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 1, 2, 3 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά ε, αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι 5 και οι 6 ταυτόσημες, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 ε, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ κατά ε, απορρίπτεται. Η 14 υπέρ ναι, κατά ε, αποχές απορρίπτεται. Και πάμε τώρα στην 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 18, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 19, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η 20-20, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του Άουτολα Κυρνίσεν υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ε, θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο, πολύ ωραία. Ε, ε ψηφίζουμε λοιπόν, ξεκινά ηλεκτρονική ψηφορία για την ε, 35. Τώρα μόνο ένας ξέχασε να ψηφίσει. 59 υπέρ, 17 υπέρ, 50 κατά. Έκλεισε η ψηφορία, αλλά πέστε μου παρόλα αυτά. Κυρία Άουταλα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι τα μέλη γνωρίζουν την τελευταία εκδοχή αυτής της τροπολογίας, διότι γίνεται πολύ πιο ακριβή η διατύπωση από τον συνάδελφο Μπρόκ και το έχω μπροστά μου. Δεν ξέρω τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Ε, θα μου επιτρέψετε να αναγνώσω την τροπολογία. Ωραία. Προτείνει συνεπώς. Προτείνει συνεπώς να αναβληθεί η διαδικασία έγκρισης της ε, Συμφωνίας Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης στην Ολομέλεια με το Τουρκμενιστάν όπως ε, σχεδιάζεται για το Μάιο και ζητά από την Κομισιόν να αναφέρει στο Κοινοβούλιο στις αρχές ε, του μηνός αυτού για τις επιπτώσεις ε, που έχει η ενδιάμεση συμφωνία στις σχέσεις με τον Τουρκμενιστάν μετά τη θέση σε ισχύ των, της συμφωνίας έτσι όπως αποφασίστηκε από το Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2008 και το αργότερο στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Bene, sì, Πολύ ωραία λοιπόν. Αυτό είναι το καθοριστικό σημείο. Μέσα στην Ολομέλεια του ε, Ιουνίου. Να, ψηφίστε, να προσθέσετε λοιπόν και αυτό ε, στον κατάλογο ψήφου. Ευχαριστώ. Όπως διάβασε και η κυρία Χάουτολα, έτσι είναι και στον κατάλογο ψηφοφοριών και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να εκφραστούμε γνωρίζοντας πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Allora, possiamo passare... Πολύ ωραία λοιπόν, μπορούμε να ψηφίσουμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία για την έκθεση. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία, παρακαλώ. Θέλετε τώρα να λάβετε το λόγο. Πρόεδρε, συγγνώμη. Ως αποτέλεσμα αυτής της ανάγνωσης κάποιοι έχουν αλλάξει γνώμη και θέλουν να ξαναψηφίσουμε, διότι έχουμε την αίσθηση ότι δεν ψηφίσαμε ε, σωστά. Ωραία. Ε, Ξεκαθαρίσαμε ότι το κείμενο το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο ψήφου με τη διευκρίνηση της κυρίας Άουτολα που προέβλεπε ένα χρονικό περιθώριο, δηλαδή μέσα στην Ολομέλεια του Ιουνίου, αυτό το ήξεραν όσοι ψήφισαν. Δεν νομίζω ότι άλλαξε τίποτα. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ο κύριος Μπροκ παρακαλώ. Δεν μας είχε υποβληθεί αυτό το χρονικό περιθώριο. Εγώ δεν ψήφισα για την έκθεση Hotel όπως ε, έχει διαμορφωθεί ή διατυπωθεί γιατί θα μπορούσε να μετατεθεί ε, ή να αναβληθεί για το διενεκές. Αλλά με την ε, χρονική προθεσμία αυτό παίζει ρόλο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή διαδικασία να πάει το ταξίδι επιτροπή να επανέλθει. Σωστή αυτή η προθεσμία. Σήμερα λοιπόν συμφωνούμε με την έκθεση αυτή και έτσι δίνουμε ένα μήνυμα ότι επιθυμούμε να είμαστε ε, επικοδομητικοί. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια δίκαιη και καλή συμβαστική πρόταση. Άρα δηλαδή κύριε Μπρόκ τι προτείνετε. Προτείνετε να ξαναψηφίσετε για την τροπολογία με αυτή την προστίκη της προθεσμίας. Μάλιστα λέει ο κύριος Μπρόκ με την προθεσμία. Πολύ ωραία λοιπόν. Αν ε, συμφωνείτε ε, με αυτή την ε, προστίκη να ξαναψηφίσουμε για την τροπολογία υπαριθμών 35 όπως διατυπώθηκε με την προστίκη χρονικού περιορισμού δηλαδή μέχρι την Ολομέλεια του Ιουνίου. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 35. Υπάρχουν ακόμα πολλοί συνάδελφοι που δεν έχουν ψηφίσει, παρότι έχουν ε, τοποθετήσει στη σχισμή τις ε, κάρτες τους. Και οι φιλελεύθεροι ε, έχουν μία ψήφο που περισσεύει. Τέλος πάντων, κλείνουμε τώρα την ψηφοφορία. Λοιπόν, 32 κατά 36 υπέρ και μία αποχή. Τώρα, τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λείπουν ακόμα συνάδελφοι, αλλά βλέπω ότι δεν θέλουν να ψηφίσουν. Α κλείσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. 59 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια ε, στον εισηγητή. Εγκρίνεται το ψήφισμα, η πρόταση ψηφίσματος. Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Μία ψηφοφορία για ένα κείμενο. Υπέρ παρακαλώ. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. άρχεται η ψηφοφορία. me Eh. Υπάρχουν nove persone che non votano μην ψηφίζουν. Λοιπόν, κλείνουμε την ψηφοφορία. 56 favorevoli. 56 ε, υπέρ, ε, μία ψήφος κατά, μία αποχή, συγχαρητήρια στις εισηγήτριες. Μην ξεχνάτε να βγάλετε, μην ξεχάσετε να βγάλετε τις κάρτες σας από τη σχισμή. Κλείσανε οι ψηφορίες, τελειώσαμε με τις ε, ψηφοφορίες.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 Bene, colleghi, per favore, vogliate prendere posto. καθίστε συνάδελφοι. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και έχουμε ιδιαίτερα φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ καθίστε. Όποιος είναι να φύγει, να φύγει γρήγορα παρακαλώ. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε τη συνέχεια των εργασιών μας. Σας παρακαλώ πολύ, Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τον Υπουργό Μαρτονή. Όπως ξέρετε, ως ΑΦΕΤ χαιρόμαστε που έχουμε μαζί μας, μεταξύ μας, τον Υπουργό Εξωτερικών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ουγγαρία έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα προς τα εμπρός με την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ και συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή μας προωθεί έναν σημαντικό διάλογο με την εκπεριτροπής Προεδρία και μέσα στα πλαίσια της ΑΦΕΤ θέλουμε να συντονίσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διεύρυνση. Γι' αυτό θα θέλαμε να μάθουμε τις προοπτικές προσχώρησης της Κροατίας. Μόλις έχουμε εγκρίνει ένα ψήφισμα για τη μελλοντική προσχώρηση της Κροατίας, γι' αυτό θα θέλαμε να μάθουμε πώς έχουν τα πράγματα στα πλαίσια της διεύρυνσης και επίσης να μας πει ο Υπουργός ε, τι συμβαίνει και στην Αλβανία μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Για να κάνει Ναι, νομίζω ότι το ζήτησα ήδη. Και εν πάση περιπτώσει όταν λάβει το λόγο ο Υπουργός νομίζω ότι θα επικρατήσει ησυχία στην αίθουσα. Ο κύριος Πόσελτ ζήτησε το λόγο. Α, όχι, ο Υπουργός έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για την απόφαση που μόλις λάβατε. Θα διευκολύνει πάρα πολύ το έργο μου. Δεδομένου ότι φαίνεται πως υπάρχει μια απόλυτη συμφωνία μεταξύ της δικής σας απόφασης και της δικής μας θέσης. Φυσικά αναφέρομαι στο θέμα της ένταξης της ε, Κροατίας. Ε, πρόκειται για μια προτεραιότητα η οποία αναφέρθηκε επανειλημμένως, ότι δηλαδή επιθυμούμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Κροατίας πριν από τη λήξη της Ουγγρικής Προεδρίας ε, να μπορέσουμε να κλείσουμε τις διαπραγματεύσεις λοιπόν. Η υπογραφή είναι μια άλλη υπόθεση. Θα ήμασταν πολύ ευτυχείς να οργανώσουμε την τελετή υπογραφής στους φίλους μας Ε, στους φίλους μας ε, Πολωνούς. Νομίζω ε, ότι όλα αυτά αποτελούν μια πολύ καλή βάση για να συνεχιστεί η στενή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πολλές φορές έχουμε ήδη αναφέρει ότι η Ουγγρική, η Ουγγρική Προεδρία επιθυμεί να είναι μια Προεδρία φιλική προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. θα συνεργαστούμε και στο τομέα της διεύρυνσης και σε όλα τα θέματα που συνδέονται με αυτήν. Ε, ελπίζουμε δε ότι ε, όχι μόνο η Ουγγρική Προεδρία θα είναι φιλική προς το ε, κοινοβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο προς την Ουγγρική Προεδρία. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να επισημάνω εδώ. Η Ουγγρική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμφότεροι είναι υπέρ της διεύρυνσης. Κάτι το οποίο αποδεικνύει και το ψήφισμα αυτό. Τούτο δεν είναι νέο βεβαίως στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι επί ετών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε προσέδιδε ιδιαίτερη σημασία στα θέματα διεύρυνσης. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πάντοτε σαφές ότι μια θεμελιώδης αξία της ολοκλήρωσης είναι ακριβώς η ανοιχτή πολιτική. Και αυτή είναι η αρχή στην οποία βασίστηκαν οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι αναπτύχθηκαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και σιγά σιγά το όραμα αυτό έγινε πραγματικότητα. Η διαδικασία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Πρόκειται για unfinished business, όπως λέμε στα αγγλικά, δηλαδή η υπόθεση δεν έχει τελειώσει ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Και βεβαίως μπορεί να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις θέσεις των χωρών μελών. Αλλά όλοι συμφωνούμε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έτσι όπως περιγράφεται στις συνθήκες, είναι ο απότερος στόχος και είναι στόχος ε, που ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης αρκεί να πράξουν όλα όσα είναι απαραίτητα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα επίσης να πω δύο λόγια σχετικά με τα δύο μέλη του, της τριάδας που προηγήθηκαν και που κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια. Αναφέρομαι στην Βελγική Προεδρία και την Ισπανική Προεδρία. Εμείς είμαστε το τελευταίο μέλος αυτής της τριάδας. Συνεχίζουμε λοιπόν το έργο το οποίο ξεκίνησαν οι άλλες δύο χώρες όσον αφορά στην ένταξη της Κροατίας. Η ε, τελευταία συνάντηση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων στις 22 Δεκεμβρίου ήταν πολύ καρποφόρα και η Βελγική Προεδρία κατόρθωσε να κλείσει τρία κεφάλαια στις διαπραγματεύσεις αυτές με την Κροατία και τούτο είναι ένα θετικό μήνυμα ε, ως προς την ένταξη της ε, Κροατίας. Συμφωνούμε ότι η ένταξη θα πρέπει να είναι προβλέψιμη, αξιόπιστη και ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρηθούν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο τις θέσεις αυτές και εμείς ως Προεδρία δεν έχουμε παρά να ακολουθήσουμε τη γραμμή που καθορίζουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Αναφέρομαι και στην ε, σχετική διατύπωση, ότι δηλαδή η ένταξη αυτή και το πέρα των διαπραγματεύσεων ε, έχει καταστεί ορατό. Όσον αφορά τα όσα η χώρα μου έζησε από την άλλη πλευρά βεβαίως, από την άλλη ε, όχθη και υπό άλλες συνθήκες, η εμβάθυνση και η προσπάθεια ένταξης της Ευρωπαϊκής η εμβάθυνση μάλλον ή η διεύρυνση είναι το πιο σημαντικό. Εμείς στη δική μας εποχή είχαμε την άποψη ότι η διεύρυνση και η εμβάθυνση δεν αποκλείουν η μία την άλλη. Αντιθέτως, πρόκειται για τάσεις οι οποίες ενισχύουν η μία την άλλη. Αν δηλαδή μελετήσουμε το ζήτημα από την ιστορική σκοπιά, θα δούμε ότι η ιστορία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, στην ιστορία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, κάθε διεύρυνση α, ακολουθήθηκε από μια διαδικασία εμβάθυνσης. Και τούτο είναι εξίσου αληθές και τώρα, διότι έχουν αρχίσει ήδη εργασίες για την επεξεργασία των συνθήκων που κατέληξαν στη συνθήκη της Λισαβόνας και Ε, βεβαίως υπάρχουν ακόμα και άλλα ε, θέματα που πρέπει να διευθετηθούν, όχι εξαιτία της διεύρυνσης, αλλά επειδή υπάρχουν ποιοτικέ διαφορές ε, και συνδέονται μάλιστα και με την εξωτερική πολιτική. Και δεν πρόκειται για χώρες οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να εκπληρώσουν κάποιες προϋποθέσεις. Βεβαίως, τούτο είναι μέρος του παιχνιδιού. Ωστόσο, διεύρυνση ενδιαφέρει και είναι προς το συμφέρον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούμε για την οικονομία και για την ανάπτυξη, για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για την βιώσιμη αηφόρο ανάπτυξη, για την ενεργειακή ασφάλεια. Και μπορούμε αμέσως να δούμε ότι όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα και συνδέονται με την ίδια την, την διεύρυνση. Η διεύρυνση λοιπόν είναι ταυτόχρονα, μας βοηθά να, ταυτόχρονα να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είμαστε υπέρ λοιπόν της διεύρυνσης και τούτο επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι έχουμε προσκαλέσει τις υποψήφιες χώρες σε πολλές φάσεις των συνεδριάσεων του Συμβουλίου μας. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων και του καθενός ξεχωριστά να περάσει το μήνυμα ότι ως μελλοντικά μέλη η γνώμη, η γνώμη αυτών των χωρών μας είναι χρήσιμη. Έτσι λοιπόν πολλά θέματα είναι στην ημερησία διάταξη και, και για μας και για εκείνους είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τις δικές τους απόψεις. Από τη σκοπιά της ε, διαδικασίας διεύρυνσης τώρα, η ένταξη της Κροατίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Διότι η απόφαση που ελάβατε δείχνει επίσης ότι δεν αφορά μόνο στην Κροατία. Πρόκειται για ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο είναι εξίσου σημαντικό και για τις άλλες υποψήφιες χώρες ή χώρες οι οποίες επιθυμούν να ε, καταστούν υποψήφιες προς ένταξη. Και είναι ένα μήνυμα και προς αυτές. Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία ένταξης εμπεριέχει πολλές δυσκολίες και πολλές προκλήσεις. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα να είναι σαφές. Το τρένο βρίσκεται σε κίνηση. Δεν γνωρίζουμε την ταχύτητα που θα αναπτύξει και δεν γνωρίζουμε ποιος και πότε θα ανεβεί σε αυτό το τρένο. Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι πάντες μπορούν να ανεβούν σε αυτό το τρένο και το τρένο προχωρά ταυτόχρονα, διότι αυτό είναι προς το συμφέρον όλων. Νομίζω ότι η ένταξη της ε, Κροατίας εμπεριέχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο πέραν αυτού του μηνύματος ε, των, ε, της ανοιχτή αγκάλης αν θέλετε. Νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό το ότι η ένταξη της Κροατίας θα διευκολύνει την περιφερειακή συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια. Γνωρίζουμε ότι η συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια είναι πολύ σημαντική και από τη σκοπιά αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική παίζει σημαντικό ρόλο. Πρόκειται για μια πραγματικότητα, μπορούμε να την επιτύχουμε, είναι μια κινητήρια δύναμη και τούτο ε, οδηγεί στην επίτευξη των πανευρωπαϊκών μας στόχων. Ε, τώρα, μέχρι τώρα μιλούσαμε για την Κροατία. Όσον αφορά στις άλλες υποψήφιες χώρες, γνωρίζουμε ότι πολλή συζήτηση γίνεται ε, γύρω από την υποψηφιότητα της Τουρκίας, της πιθανότητες ένταξης, την έκβαση των διαπραγματεύσεων κλπ. Υπάρχουν θέματα ε, γενικότερης στρατηγικής, παγκόσμιας στρατηγικής και ακούγεται συχνά ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εξαρτάται και από το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις με κάποιες δυνάμεις. Και πρώτα απ' όλα με την Τουρκία. Δεν είναι μυστικό νομίζω ότι είμαστε μεταξύ εκείνων πιστεύουν ότι η Τουρκία έχει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει θέση μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να διαδραματίσει έναν πολύ πιο επικοδομητικό ρόλο στην παγκόσμια πολιτική σκηνή αν ολοκληρωθεί η ένταξη της Τουρκίας. Πέραν όμως της παγκόσμιας στρατηγικής ε, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τους προσεχείς ε, έξι μήνες ή πιο συγκεκριμένους προσεχείς πέντε μήνες, αν μπορούμε να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά πολιτικά ε, προβλήματα, ζητήματα, όπως επίσης και άλλα ευαίσθητα ζητήματα. Πρέπει να σημειωθεί η πρόοδο σε κάποια κεφάλαια, τους προσεχείς μήνες. Βεβαίως τούτο δεν εξαρτάται αποκλειστικά από μας. Εν πάση περιπτώσει, ε, τούτο αποτελεί τη δική μας φιλοδοξία. Ισλανδία. Είναι εντελώς διαφορετική η περίπτωση. Πρόκειται για μια χώρα ε, η οποία συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, το Σέγγεν, αλλά υπάρχουν και δυσκολίες. Πού έγκυται οι δυσκολίες. Ε, είμαστε στη φάση του screening. Το Συμβούλιο αναμένει τα αποτελέσματα αυτών των μελετών και μόλις έχουμε τα αποτελέσματα θα προχωρήσουμε στον καθορισμό τη ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων. Κατά πάσα πιθανότητα τούτο θα είναι προς το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας τον Ιούνιο. Και νομίζω ότι κατόπιν θα είναι δυνατόν να συζητήσουμε θέματα που θεωρούνται πιο δύσκολα και τα οποία θα επιληθούν ε, σε συνεννόηση με τα δύο μέρη. Ε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες σχετικά με τις σχέσεις μας με άλλες χώρες της περιοχής. Γνωρίζετε ότι έχουμε προβλήματα και γνωρίζετε επίσης και τα στοιχεία εκείνα τα οποία αποτελούν ε, πρόσκομα, εμπόδιο για την πρόοδο των σχέσεων. Ε, τούτο ισχύει και για τη Φιρόμ, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εμείς προτρέπουμε τα μέρη να επιλύσουν το πρόβλημα του ονόματος και μόλις επιληθεί το ζήτημα της ονομασίας δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Επίσης, ε, με μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε και το Μαυροβούνιο, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου. Έχουν τεθεί επτά προϋποθέσεις, επτά όροι. Ε, που πρέπει η χώρα αυτή να εκπληρώσει για να ξεκινήσει και με αυτήν η διαδικασία ε, των διαπραγματεύσεων. Υπήρχαν βεβαίως δυσκολίες και ανησυχίες στο παρελθόν, αλλά και σήμερα. Ε, ε του, τούτο έρχεται, μάλλον η σεπήρωση του ε, ήρθαν τα γεγονότα ε, των τελευταίων ημερών στην Αλβανία δεν έχει βέβαια άμεση σχέση με την διεύρυνση, ωστόσο όλα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, γι' αυτό και παρακολουθούμε πολύ στενά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις ε, στη χώρα αυτή. Η Προεδρία δεν θέλει να λάβει θέση ε, σε μια πολιτική συζήτηση. Θέλουμε να προτρέψουμε όλες τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταλήξουν σε ένα μόντους βιβέντη. Σε μια λύση συγκατοίκησης που θα επιτρέψει να γίνουν βήματα προς την κατεύθυνση της ε, ένταξης σε ευρωπαϊκές δομές. Η εξωτερική υπηρεσία δράσης κάνει τα απαραίτητα στον τομέα αυτό. Σήμερα έγιναν σημαντικές συναντήσεις με σκοπό να προτρέψουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν μεταξύ τους. Είναι υποχρέωσή μας να λειτουργήσουμε ως διευκολυντές, όχι ως αυτοί που θα επιλύσουν τα προβλήματα. Γενικά θα ήθελα για μία ακόμη φορά να επαναλάβω ότι βασιζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο που είναι υπέρ της διεύρυνσης, εμείς δε σε επίπεδο συμβολίου θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Καθορίζοντας τους στόχους μας, για κάθε υποψήφιο θα θέλαμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Ίσως τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Ας πούμε στην περίπτωση της Σερβίας, η σερβική πλευρά θα μας υποβάλει την απάντηση σε ένα ερωτηματολόγιο που έχει τεθεί και με βάση αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατυπώσει τη δική της γνώμη. Διαφορετικά θα είναι τα βήματα με τις άλλες χώρες. Αλλά αυτό που επιθυμούμε είναι να σημειωθεί πρόοδος για κάθε μία από τις χώρες. Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε ανοιχτοί, ότι είμαστε αξιόπιστοι. Τονίζουμε ότι όλοι θα πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν και θέλουμε ταυτόχρονα να αποδείξουμε ότι η διαδικασία της διεύρυνσης και το, της ένταξης ε, δεν έχει κλείσει. Θέλουμε, ε, θέλουμε μια διαρκώς ανοιχτή ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ξεκινάμε με τη συζήτησή μας. Δυστυχώς στις 5 πρέπει να κλείσουμε διότι ο Υπουργός έχει μία άλλη δέσμευση και εμείς θα έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο Φίλε. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που ζήτησαν το λόγο, άρα είμαι υποχρεωμένος δυστυχώς να σας επιβάλλω να μιλήσετε για ένα λεπτό και μόνο. Εάν τα καταφέρετε ο κύριος Σαλαφράγκα, καλωσορίσατε. Είπατε ότι θέλετε, κύριε Υπουργέ, να είσαστε φίλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Ε, ένας φίλος θα πρέπει να ακούει και δυσάρεστα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι θα σας υποστηρίξουμε μέσα στα πλαίσια της ε, Προεδρίας. Πέρα από την έκθεση Σβόμποτα για την κατάσταση στην Κροατία δεν πιστεύετε ότι υπάρχει μία κόποση στη διαδικασία προσχώρησης τη στιγμή που ζούμε μία χρηματοπιστωτική κρίση, ζούμε μία κατάσταση σαν τον μύθο του Ναρκίσου. Δηλαδή, προβαίνουμε σε μία πράξη αυταρέσκειας. Το θέμα της διεύρυνσης πώς θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε, διότι έχουμε προβάλλει μία πρόταση συμβιβασμού και δεν θα ήταν σκόπιμο να συσταθεί μία task force η οποία να παρακολουθεί τη διαδικασία διεύρυνσης μέσα στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών. Τα καταφέρατε κύριε Σαλαφράνκα. Ο συνήθως, ο κύριος Σεβερίν. Ευχαριστώ. Γνωριζόμαστε εδώ και μακρύ χρονικό διάστημα, κύριε Υπουργέ, κύριε ε, Ματώνη. Αλλά έμαθα ότι γεννηθήκατε στο Κόλες Βάρες και εγώ ως Ρουμάνος σοβουνιστής θα πρέπει να τονίσω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με εξέπληξε ιδιαίτερα. Εν πάση περιπτώσει, περνώντας σε πιο σοβαρά θέματα ελπίζω να δράσετε έτσι ώστε να άρουμε ε, μία προκατάληψη, διότι η διεύρυνση θεωρήθηκε φόρτος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να τα καταφέρετε αυτά, αυτό εξ ονόματος της Προεδρίας. Δηλαδή η διεύρυνση δεν είναι άχθος. Δεύτερον, Έχουμε μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με δύο στρατηγικούς εταίρους, δηλαδή της ΗΠΑ και τη Ρωσία. Θα ήθελα λοιπόν, απαντώντας, να μας μιλήσατε για το πώς η Ουγγρική Προεδρία προσεγγίζει το θέμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ ημών και της Ρωσίας διότι σήμερα μιλήσαμε με εκπροσώπους της Ρωσίας και φαίνεται ότι το θέμα αυτό έχει μεγάλη σημασία και για εκείνους και για μας. Ο κύριος Κάτσιν, συγητής για τη διεύρυνση προς τη Σερβία. Ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. I would like to welcome... Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, αλλά όπως γνωρίζετε έχετε τις δικές σας προτεραιότητες και η ζωή συνεχίζεται μέσα στη δυναμική της. Τα γεγονότα στα τύρανα μας εξέπληξαν όλους και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να δράσουμε επιχειρησιακά. Ήταν έκπληξη και για την Προεδρία αυτή η μεγάλη κλειδονισμή, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Θα πρέπει να πείσουμε και τον Πρωθυπουργό και τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης να είναι πιο ειλικρινής και πιο όρημοι, πιο ενήλικοι αν θα μπορούσα να πω, πιο ενήλικες. Ναι, Αναφέρθηκα και στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, αλλά δυστυχώς ε, έτσι έχουν τα πράγματα. Θα ήθελα εσείς να ερμηνεύσετε τα πρόσφατα γεγονότα και να μας πείτε ποιες είναι οι προβλέψεις σας. Ευχαριστούμε κύριε Κατσίν. Μπραντνερ, για ένα λεπτό. thank you very much. I have just two quick questions. One... Δύο ερωτήσεις σε σχέση με την Αλβανία κατά πόσο ε, έχετε κάποιο πρόγραμμα, κάποιο σχέδιο, πώς θα δράσετε, διότι οι δύο δυνάμεις πρέπει να συνεπάρξουν. Και αυτό το είδαμε και στα πλαίσια του ΟΑΣΕ. Ίσως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι προτίθεστε να κάνετε. Και το δεύτερο ερώτημα, εξ ονόματος κυρίας Λούνατσεκ, ως προς το κοσυφοπέδιο κατά πόσο θα ξεκινήσετε έναν διάλογο για το καθεστώς των θεωρήσεων. Ευχαριστούμε την κυρία Μπραντνερ. Ο κύριος Άτκινς, ο επικεφαλής των συντηρητικών. Εντάχει. Μόλις επανήλθα από τη Μέση Ανατολή και μέσα στο εξάμεινό σας, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να δείτε πώς δαπανώνται τα κονδύλια μέσα στα πλαίσια της ε, δράσης του κουαρτέτου που καταλαμβάνει μία σουίτα σε ένα ακριβό ξενοδοχείο της Ιερουσαλήμ. Όποια θέση και να λάβετε επί του θέματος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κουαρτέτο είναι μία κατασπατάληση χρημάτων, δεν καταφέρνει σχεδόν τίποτα και στο Συμβούλιο ίσως θα ήταν σκόπιμο να δούμε πώς δαπανούνται τα χρήματα των φορολογουμένων και κατά πόσο ε, φτάνουν σε, καλά χέρια. Και εδώ αναφέρομαι στον κύριο Μπλερ ιδιαίτερα, ο οποίος πιστεύω ότι δεν καταφέρνει τίποτα. Κόντις, εισηγητής για θέματα Αλβανίας. Ο κύριος Χουντής, με συγχωρείτε. Επειδή ο χρόνος είναι σύντομος, δεν θα ήθελα να σχολιάσω τις μετριοπαθείς εκτιμήσει του Υπουργού σε σχέση με το θέμα της διεύρυνση και θα ήθελα να πω δύο κουβέντε για το θέμα της Αλβανίας. Νομίζω ότι πρέπει να εκφράσουμε τη θλίψη μας για το θάνατο και το τραυματισμό ανθρώπων που διαδήλωναν στην Αλβανία. Νομίζω ότι πρέπει να εκφράσουμε την απέτησή μας να, αποδοθεί δικαιοσύνη σε σχέση με τι αιτίε και τους υπεύθυνου αυτών των θανάτων και των τραυματισμών, χωρίς παρεμβάσεις διαφόρου τύπου που δυσκολεύουν την απόδοση δικαιοσύνη. Όσο αφορά αυτά καθ' αυτά τα γεγονότα, θέλω να σα πω ότι από μια άποψη, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ήταν και τόσο απρόσμενα, Καθώ είχαμε ένα πολιτικό αδιέξοδο που δεν βρισκόταν λύση εδώ και 1,5 χρόνο, ενώ, όπως ξέρετε, η αφορμή ήταν ένα φαινόμενο ακόμα δωροδοκίας και διαπλοκής, που όπως είχαμε διαπιστώσει στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε πάρει τέτοια έκταση που εμπόδιζε να λυθούν μια σειρά προβλήματα. Το ερώτημα λοιπόν, ναι κύριε Πρόεδρε, είναι από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Προφανώς δεν πρέπει να μείνουμε αδρανείς, ενδεχομένως να τεθεί το θέμα στην έκτακτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συζητηθεί εκεί. Εκτιμώ τη μετριοπαθή στάση της Προεδρίας ότι όποια παρέμβαση γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι προσεκτική, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να βοηθήσουμε τι πολιτικέ δυνάμει να αντιληφθούν ότι με ευθύνη και οριμότητα πρέπει να λύσουν το, πολιτικό πρόβλημα και τα άλλα προβλήματα τη Αλβανία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χούντι, ο κύριο ε, Κούκαν, που είναι πρόεδρος ε, της ε, αντιπροσωπείας με τις χώρε των Ανατολικής Ευρώπης. Και εσείς λυπάμαι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, σας καλωσορίζουμε κύριε Υπουργέ, κύριε Μάρτονη. Ε, σας συγχαίρουμε για τις προτεραιότητες που έχει ορίσει η Ουγγρική Προεδρία. Σωστά έχουν οριστεί. Εγώ ε, χαίρομαι ιδιαίτερα πώς προτεραιότητα συμπεριλάβατε και τη διεύρυνση. Όσον αφορά στην Αλβανία, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Μας ανησυχεί τα μάλα και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί, ότι θα υπάρξει φως ίσως στο τέλος του τούνελ. Μα εγώ ούτε καν τούνελ δεν βλέπω. Εκείνο λοιπόν που χρειαζόμαστε τώρα <clears throat> είναι όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να στείλουν ένα κοινό ισχυρό μήνυμα προς όλες τις διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα μήνυμα όπου θα καλούνται οι πολιτικοί ηγέτες στην Αλβανία, να συμπεριφέρονται ως μέλη του ΝΑΤΟ και ως μελλοντικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε και να στέλνουμε ε, μηνύματα μέσα από διαφορετικά κανάλια και σε διαφορετικές διευθύνσεις δεν θα βοηθήσουμε, θα υπάρξει κλιμάκωση της κατάστασης. Ε, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ένα και ισχυρό μήνυμα. Και εσείς ξέρετε μπορείτε να παίξετε ρόλο στο να γίνει κάτι τέτοιο. Πολύ ωραίο λέει Πρόεδρος, ε, η κυρία Μίνιθ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα μας μιλήσετε για τις προτεραιότητες ως προς την διεύρυνση. Ελπίζω να μας μιλήσετε και για άλλα θέματα εξίσου σημαντικά της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αφορούν την διεύρυνση που αφορά την ε, τρόικα των προεδριών σε σχέση με προτεραιότητες, ενδεχόμενες προτεραιότητες, έτσι ώστε να δώσουμε συνέχεια στην ε, διάσκεψη κορυφής ε, Ιβηρικής, Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη και τις σχέσεις με το Μερκοσούρ. Ελπίζω να μπορέσετε σε άλλη περίσταση να μας μιλήσετε για αυτές τις προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Κύριε ε, που σεβάστηκε το χρόνο που τη διατέθηκε. Ο κύριος Σούλτς παρακαλώ για ένα λεπτό. Ε, κύριε Υπουργέ, ε, πολύ σωστά επισημάνατε την εκπλήρωση των κριτηρίων της ε, Κοπενχάγης από πλευράς ε, μελλοντικών υποψηφίων χωρών. Όμως τι γίνεται με την τήρηση των κριτηρίων αυτών όσον αφορά στα νυν κράτη-μέλη και εδώ λυπάμαι, αλλά εσείς δίνετε ένα πολύ κακό παράδειγμα κακό παράδειγμα και κυρίως σε σχέση με την άμπλυνση των κριτηρίων. Ε, σήμερα ακούσαμε τον Ρώσο πρέσβη, τον κύριο Τσίχοφ, ο οποίος ε, όσον αφορά στην έλλειψη ελευθεροτυπίας ε, στην Ρωσία μας είπε ασχολείται με τα δικά σας και μας παρέπεμψε ε, σε εσά στην Ουγγαρία το ίδιο ακούμε και από την ε, Λευκορωσία και από την Ουκρανία. Σε λίγο και από την Αλβανία θα τα ακούσουμε αυτά. Εσείς λοιπόν πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτές τις ε, καταγγελίες. Ευχαριστούμε. Ε, Σοπφιν, ένα λεπτό. Σας καλωσορίζουμε θερμά στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αναφερθήκατε στην Τουρκία η Τουρκία όλο και περισσότερο υιοθετεί μια πολύ ισχυρή θέση μέσα στην περιοχή και νομίζω ότι παίζει ένα όλο και πιο σημαντικό ρόλο ε, στο, σε σχέση με το Ιράν, τον Κάφκασο και την Μέση Ανατολή. Εσείς τι πιστεύετε για αυτό τον πολύ ισχυρό ρόλο που αναλαμβάνει η Τουρκία στην περιοχή. Ευχαριστούμε. Αρλάκι, Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που είπατε για την Τουρκία. Βλέπω ότι η Ουγγρική ε, Προεδρία προτίθεται να ασχοληθεί περισσότερο με τη διεύρυνση και να έρθει πιο κοντά στο μεγάλο μας γείτονα. Τώρα, τι έχετε συγκεκριμένα κατά νου, έτσι ώστε αυτές τις προθέσεις σας απέναντι στην Τουρκία να τις μετατρέψετε σε συγκεκριμένες πράξεις κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά την Αλβανία, η οποία επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις όμως είδαμε την αστυνομία στην Αλβανία να πυροβολεί κατά διαδηλωτών. Σκοτώθηκαν άνθρωποι Εντάξει, υπήρξε ε, αμέσως, ε, ευθύς αμέσως μετά τα γεγονότα αυτά μια ενθαρρυντική αντίδραση της ε, δικαστικής εξουσίας στην Ουλβανία. Εγώ ρωτώ λοιπόν, εσείς τι πιστεύετε, πώς μπορεί να ενισχυθεί η δικαστική εξουσία στην Αλβανία και πώς μπορούμε να πείσουμε την αστυνομία στην Αλβανία να σέβεται τις προδιαγραφές και τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόκβιλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η δική μου ερώτηση αφορά τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, ακόμα και αν δεν είναι θέμα διεύρυνσης, διότι πριν από λίγες μόνο ε, ημέρες η ύπατη εκπρόσωπος είπε στα μέσα ότι συζητιέται ε, να αρθεί το εμπάργο όπλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Κίνας. Το Κοινοβούλιο όμως έχει πει να γίνει κάτι τέτοιο μόνο εφόσον υπάρξει κάποια διαλεύκανση της υπόθεσης των θυμάτων της Τιαναμέν της πλατείας. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολεί στους επόμενους έξι μήνες και ποια είναι η δική σας η θέση επί του θέματος. Πρέντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισήγησή σας. Διαπίστωσα με μεγάλη χαρά ότι σε ένα έγγραφο που ορίζει τις προτεραιότητες για τη διεύρυνση αναφέρεται ότι θα ανοίξετε το πρώτο κεφάλαιο για την προσχώρηση της, Ιρλα... της Ισλανδίας. Γνωρίζοντας πόσο λεπτό είναι το θέμα της κοινή γνώμης στην Ισλανδία, θεωρείτε ότι θα πρέπει να ανοίξετε καταρχήν τα δύσκολα κεφάλαια ή τα πιο εύκολα κεφάλαια για την μελλοντική προσχώρηση. Ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Μπόσκουρτ για ένα λεπτό. Κύριε ε, Υπουργέ, στα εισαγωγικά σας λόγια είπατε ότι η Ουγγαρία τάσεται υπέρ της διεύρυνσης και είπατε ότι θα θέλατε να ανοίξετε περισσότερα κεφάλαια με την Τουρκία τους επόμενους μήνες τα πράγματα ε, ακολούθησαν ε, μία δύσκολη οδό και αδιέξοδα από τις στάση ορισμένων κρατών μελών. Τι θα κάνετε έτσι ώστε να κινηθεί εκ νέου η διαδικασία. Γιατί παραμένουν πολλά κεφάλαια. Ως προς την Κροατία μιλάμε για την διεύρυνση η οποία θα οδηγήσει και στη ε, διεύνηση προς τα, τα άλλα Δυτικά Βαλκάνια. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει με το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Τάνοκ για ένα λεπτό. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Υπουργό μια ερώτηση γενικής υφής. Ποιος είναι ο ρόλος της εκπεριτροπής Προεδρίας του Υπουργού Εξωτερικών σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και τη διεύρυνση, διότι έχουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πλέον και τον ειδικό ρόλο της ύπατης εκπροσώπου. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σκόπιμο να σας απευθύνουμε το λόγο ως προεδρεύοντα. Βρισκόμαστε σε μία ε, γκρίζα ζώνη. Είσαστε πρώτος μεταξύ ίσων μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών στο Συμβούλιο ή κάτι τέτοιο δεν θα ισχύσει τους επόμενους μήνες. Ως προς τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια, εγώ είμαι εισηγητής για το Μαυροβούνιο. Θα γίνουν συζητήσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα και υπάρχει και η έκθεση Dick Marty η οποία καταφέρεται κατά του κοσυφοπεδίου όπου υπάρχει οργανωμένο έγκλημα και λαθρεμπόριο, διακίνηση ναρκωτικών. Τι μπορείτε να κάνετε αν λάβετε υπόψη ότι εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τη Σερβία επειδή υπάρχει μεγάλη μειοψηφία στη Βοηβοδίνα. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Το λόγο έχει ο κύριος Πόσελτ για ένα λεπτό. Έχω τρεις ε, πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτον, ε, σας συγχαίρω ε, για αυτά που είπατε για την Κροατία. Εμείς επιθυμούμε οι διαπραγματεύσεις να ε, ολοκληρωθούν υπό την Ουγγρική Προεδρία έτσι ώστε το φθινόπωρο να ψηφίσουμε επιτέλους για την Κροατία και του χρόνου τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην επικύρωση. Δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω μετά κατά πόσον υπάρχει ε, ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων με την Δημοκρατία της Μακεδονίας. Γιατί και εκεί ελπίζουμε σύντομα να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία. Και το τρίτο που θέλω να πω, στη Σερβία υπήρξαν κατεδίκες ε, σε κάποια περίεργη δίκη Αλβανών και Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε ένα από τα καλύτερα δίκαια προστασίας ε, μειονοτήτων στην Ευρώπη. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, την Σερβία θα πρέπει να την μελετήσετε και κάτω από αυτό το πρίσμα της προστασίας των μειονοτήτων. Κράιστοφλα για ένα λεπτό. Και εγώ θα ήθελα να σας καλήσω θερμά κύριε Υπουργέ και χαίρομαι που θέλετε να συνεργαστείτε με εμά σε φιλικό πνεύμα. Και εγώ το θέλω αυτό και το θεωρώ και αυτονόητο. Βεβαίω είναι σαφέ ότι στα κοινοβούλια πρέπει κανεί να μιλάει και επί τη ουσία. Σα παρακαλώ λοιπόν όταν ασκούμε κριτική να μην θεωρείτε ότι υπάρχει αντιπάθεια προς τον ουγγρικό λαό, απλά διαφωνούμε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Και ρωτώ, αυτό το αδιέξοδο που διαπιστώνω με την Τουρκία στις ε, διαπραγματεύσεις ε, ε, και οφείλεται στο Κυπριακό, η Τουρκία θα πρέπει ίσως να τηρήσει τις συνθήκες οι οποίες έχουν υπογραφεί εδώ και αρκετό καιρό. Έτσι δεν είναι. Πέταρλε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Υπουργό και τον συγχαίρω που έχει αναλάβει και πάλι τα καθήκοντα του Υπουργού. Το εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του. Ένα έργο πολύ σημαντικό να αφορά την διεύρυνση και ε, αυτό και σε σχέση με τις αντιδράσεις των ευρωπαϊκών οργάνων. Η ερώτησή μου βλέπετε να υπάρχουν εμπόδια κόμματα στα κεφάλαια της ενέργειας και τι πρόκειται να κάνετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Πολύ ωραία λοιπόν. Ολοκληρώνω κύριε κύριος ο οποίος ήταν την πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Υπουργέ, ως ε, Ούγγρος από τη Ρουμανία χαίρομαι που έχουμε την Ουγγρική Προεδρία και νομίζω ότι εσείς ε, μπορείτε να εκπροσωπήσετε τα συμφέροντα της Ουγγαρίας. Η Ρουμανία είναι στο Σέγκεν και υπάρχει στρατηγική για τις περιοχές του Δουνάβου, του Δούναβη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να εξεταστούν και πρέπει να δούμε και ε, το θέμα του εικονικού σιδηρού παραπετάσματος. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μία εμβάθυνση σε θέματα διεύρυνσης. Είναι σημαντική η προσχώρηση των Βαλκανικών ε, κρατών, την εταιρική σχέση με τις ε, ανατολικές χώρες, η Ουκρανία και η Μολδαβία πρέπει και αυτές να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως μπορείτε εσείς να προωθήσετε το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. 19 ε, ερωτήσεις, ε, μάλλον 19 παρεμβάσεις, περίπου 25 ερωτήσεις και έχετε ένα τέταρτο για να απαντήσετε. Ε, μάλλον Ηράκλειο το έργο σας. Ας δούμε τι θα καταφέρετε. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος και γοργός στο μέτρο του δυνατού. Ε, δεν θα κάνω χρήση της μητρικής μου γλώσσας για να διευκολύνω το έργο των διερμενέων. Ακόμα και στα θέματα τα ουγγρικά θα απαντήσω στην Εσπεράντο. Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως. Έθεσε ο κύριος Αλαφράγκα το θέμα ότι υπάρχει μία κόπωση διεύρυνσης. Ε, δεν είναι απλώς κόπωση κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πιο βαρύ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λοιπόν προσπαθούμε να τονίσουμε ότι είναι και προς το δικό μας συμφέρον. Υπό την παρούσα κατάσταση της πορεί αργής ανάκαμψης από την χρηματοοικονομική κρίση, οι πάντες κατανοούν ότι η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, η διεύρυνση των αγορών γενικότερα, η διασφάλιση της ενέργειας, της προμήθειας ενέργειας και η αύξηση της περιφερειακής συνεργασίας είναι πράγματι υπέρ των δικών μας συμφερόντων, είναι προς το συμφέρον μας. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στην επικοινωνία μας. Όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, όχι, αλλά επειδή έχουμε πραγματικά απτά οικονομικά συμφέροντα. Και δεν ομιλώ βέβαια για την προβολή των αρχών και αξιών μας. Τώρα, την Ισία. Υπήρξε η ιδέα άμεσων επισκέψεων στη χώρα αυτή. Η αντίδραση ήταν ότι θα ήταν πολύ πρόωρο υπό το φως της κατάστασης που επικρατεί εκεί. Για να συνομιλήσει κανείς με ανθρώπους εκεί χρειάζεται συνομιλητή και ακόμα το σκηνικό δεν είναι απολύτως σαφές ποιοι θα είναι οι συνομιλητές. Αυτό που θα ήθελα απλώς να επισημάνω είναι ότι η κατάσταση είναι μεταβατική, πάρα πολύ μεταβατική. Κάποιοι ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις, κάποιοι μιλούσαν για την επανάσταση, την επανάσταση των γεσεμιών, αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις από κοντά, να παρακολουθήσουμε επίσης από κοντά τις επιπτώσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχει άμεσο συμφέρον, ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την παρούσα στιγμή νομίζω ότι οποιοδήποτε συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει να εξεταστεί προηγουμένως πολύ προσεκτικά. Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν επισκέψεις ή δεν θα γίνουν επισκέψεις είτε ομάδων μιας ομάδας της αποστολής είτε υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή. Θέλουμε να βοηθήσουμε διότι είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι αλλά το θέμα απαιτεί περισσότερη συζήτηση και ε, μελέτη για να μπορέσουμε να καταλήξουμε καταρχήν σε κάποια συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουμε υπό την παρούσα κατάσταση. Και πάλι επαναλαμβάνω το επιχείρημά μου ότι ναι, η διεύρυνση δεν είναι βάρος. Δεν είναι άχθος. Είναι και προς το δικό μας συμφέρον. Τώρα, σχετικά με τις στρατηγικές μας σχέσεις, Ηνωμένε Πολιτείε. Σύντομα συζητήσαμε το θέμα αυτό στο πλαίσιο της συζήτηση για το εξωτερικό εμπόριο και πάλι θα έρθω στο ε, αγαπημένο μου θέμα που είναι το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο. Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχει ενδιαφέρον μεταξύ των χωρών μελών. Συμφωνήσαμε επίσης ότι αναφέρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως στρατηγικό εταίρο και μερικές φορές το σμπερδεύουμε και με άλλους στρατηγικούς εταίρους που είναι εξίσου σημαντικοί. Αλλά πιστεύουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι απλό στρατηγικό εταίρο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο φυσικό μα σύμμαχο. Και τούτο σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε σε σημαντικό βαθμό και την οικονομική διάσταση, όπως και την κανονιστική διάσταση των σχέσεών μας. Αυτό θα δώσει νέα όθηση, νέα ορμή ε, στην ενίσχυση του διατλαντικού κρίκου, της σχέσης. Η Ρωσία αναφέρθηκε επίσης στο πλαίσιο της συζήτησης για το εξωτερικό εμπόριο. Ο πρόεδρος, μάλλον η Προεδρία, συγγνώμη, υποστηρίζει ενεργά την ένταξη της ε, Ρωσίας στο Παγκόσμιο Οργάνωση Εμπορίου, στον ΠΟΗ, διότι θα Εποφεληθεί βεβαίως η Ρωσία από την ένταξη, ενώ ταυτόχρονα θα ε, ε, υποχρεωθεί να τηρήσει όλους τους κανόνες και τους όρους που προκύπτουν από αυτήν. Έρχομαι τώρα στην Αλβανία. Συμφωνώ απόλυτα ότι η ζωή έχει τη δική της δυναμική. Τούτο έχει αποδειχθεί πολλές φορές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε το βέλτιστο δυνατό. Πώς δηλαδή μπορούν να συμφιλειωθούν οι δύο πλευρές. Και ε, όταν συνέβη αυτό υπήρξαν, υπήρξε μια καρποφόρα συζήτηση και οι δύο πλευρές θέλησαν δεσμεύτηκαν να καταβάλουν προσπάθεια για να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι προφανές όμως ότι τούτο δεν συνέβη. Ναι λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Αλλά ένα πράγμα που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε συμπεριφορές στα μέρη μπορούμε να τους ενθαρρύνουμε, μπορούμε να τους εξηγήσουμε ότι αν συνεχίσουν ε, αυτή την ε, συμπεριφορά θα χάσουν την ευρωπαϊκή προοπτική και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα και ελπίζουμε ότι θα καταλάβουν αυτό το μήνυμα. Επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε τον αλβανικό λαό που το αξίζει. Αυτό όμως που δεν θέλω να κάνουμε είναι να πάμε με το μέρος του ενός ή του άλλου σε αυτή την πολιτική διαμάχη την εσωτερική της Αλβανίας. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι εξημών με ύψιλον θα προτιμούσατε να λάβουμε θέση. Αλλά ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε, όχι εξαιτία του ρόλου μου, αλλά επειδή πιστεύω ότι δεν θα είναι και πολύ βοηθητικό. Πρέπει να, να τηρηθούν οι βασικοί κανόνες. Ε, εν τω μεταξύ πρέπει να πω ότι διεξάγονται ήδη έρευνες για τα αίτια, για το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια των ε, διαδηλώσεων ή ακόμα οργανώνονται ή σχεδιάζονται ε, διαδηλώσεις. Ίσως ε, η διοργάνωση μεγάλων διαδηλώσεων μπορεί να μην βοηθάει πάρα πολύ, μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερες εντάσεις κλπ. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε και τα όρια μας. Κωσυφοπαίδιο. Υπάρχει ένα ισχυρό επιχείρημα ότι το Κωσυφοπαίδιο δεν μπορεί να παραμένει ως μια μαύρη τρύπα. Πώς να το πω έτσι πολύ ευγενικά, δεν υπάρχει και μεγάλος ενθουσιασμός για διάθεση, για απελευθέρωση μάλλον του καθεστώτος ε, θεωρήσεων υπό τις σημερινές συνθήκες. Δεν έχει σημειωθεί ε, πρόοδο στο τομέα της συμφωνίας επαν... Ε, διότι εν πάση περιπτώσει πρέπει καταρχήν να ε, τηρηθούν και να εκπληρωθούν κάποια βασικά κριτήρια. Τώρα, πώς δαπανώνται τα κονδύλια, τα κεφάλαια. Με κάθε σεβασμό, νομίζω ότι το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί στην ε, εξωτερική υπηρεσία. Στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δηλαδή. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν κάνουμε δηλώσεις του τύπου μόνον πληρώνουμε, δεν είμαστε παίκτες, δεν... Στόχος μας είναι να είμαστε παίκτες. Και η άποψή μου είναι ότι στο, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων η αρρωγή, η συνεισφορά και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοια που πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο στη Μέση Ανατολή. Κάποιος αναφέρθηκε διατύπωσε μάλλον την μεγάλη ανησυχία για την Αλβανία. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να σταλεί ένα ενιαίο και συγκεκριμένο μήνυμα. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να συντονίζουμε και τα μηνύματα που στέλνουμε και τις ενέργειές μας. Αυτό είναι προς το γενικότερο συμφέρον και συνδέεται στενά με όσα αρχικά προηγουμένως συζητήσαμε ως προς τη διεύρυνση. Και εδώ τώρα έρχομαι ε, ε, ε, ενώπιό μου μπαίνει το τι εμπίπτει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και τι όχι. Περού και Κολομβία, παραδείγματο χάρη, συζητήθηκαν εχθέ στο Συμβούλιο Εξωτερικού Εμπορίου και τέθη ένα ερώτημα εκεί. Εδώ τώρα δεν είναι πολύ εύκολη η κατάσταση, διότι όπως γνωρίζετε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και όταν συζητείτε η πολιτική ε, εξωτερικού εμπορίου θα πρέπει να προεδρεύει η Προεδρία. Ενώ τα εξωτερικά ζητήματα, στα εξωτερικά ζητήματα προεδρεύει η ύπατη εκπρόσωπος. Αυτό με φέρνει στο άλλο ερώτημα. Ποιος είναι ο ρόλος μου. Να εξηγήσω το ρόλο δηλαδή της εκπεριτροπής Προεδρίας σε σχέση με την εξωτερική δράση. Νομίζω ότι δεν είναι γκρίζα τα πράγματα, σκοτεινά. Είναι όμως ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου έχει αρκετά ξεκαθαριστεί. Ε, χρειάστηκε λίγος χρόνος, αλλά η διεύρυνση ας πούμε ανήκει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Από την άλλη θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων πρέπει να είναι πιο δραστήριο στα οριζόντια θέματα και και ως προς τις συνεδριάσεις αλλά και γενικότερα στο follow-up αφού λαμβληφθούν οι αποφάσεις από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Από την άλλη, οι εξωτερικές υποθέσεις, στις εξωτερικές υποθέσεις προεδρεύει μετά τη Λισαβόνα η, η υπατή και όχι ο Υπουργός Εξωτερικών της προεδρεύουσας χώρας. το αν είμαστε πρίμους είτε πάρες ή όχι, ίσοι μεταξύ ίσων ή όχι, δεν το γνωρίζω. Αλλά μπορείς να προσκληθείς ή να σου ζητηθεί ή να αναλάβεις ειδικέ αποστολές. Πράγμα το οποίο γινόταν και πριν βεβαίως. Και ακόμα και πριν από την εκπεριτροπής Προεδρία. Παραδείγματο χάρη η ύπατη εκπρόσωπο ζήτησε από ένα μέλος του, της, Τριάδας να αναλάβει μια συγκεκριμένη αποστολή και το έπραξε. Αλλά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αυστηρά αυτά καθεαυτά, για αυτά αυτά, δεν είμαι εξουγιοντοδημένος, δεν έχω το δικαίωμα να ομιλώ εξ ονόματος της ΥΠΑ της εκπροσώπου, εκτός και αν μου ζητηθεί να το πράξω. Πράγμα που δεν έχει συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός όταν γίνονται προτάσεις, σχόλια, συστάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Και τώρα έρχομαι στο κατάλογο των ερωτήσεων. Έρχομαι στο θέμα του νόμου σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία. Θα φορέσω δηλαδή το ουγγαρέζικο καπέλο μου για ένα-δύο λεπτά. Αυτό που συνέστησα ήδη πριν από δύο-τρεις εβδομάδες, ήδη, σε εκείνους που θέλουν να κρίνουν οποιαδήποτε νομοθεσία, είπα ότι πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά και να αναλύσουν αυτή τη νομοθεσία. Το δεύτερο, που είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέγνωσε πράγματι τη νομοθεσία την, την λοιπόν την ανέλησε και ε, κατέληξε σε εντυπωσιακά και πολύ σχετικά συμπεράσματα. Άρα λοιπόν η δεύτερη σύστασή μου είναι οποιοδήποτε θέλει να κρίνει αυτό το νόμο ή ευρύτερα να ασχοληθεί με τις ελευθερίες, τη δημοκρατία κλπ. Επίσης πρέπει να διαβάσει την επιστολή του Επιτρόπου Κρόσου θα είναι πολύ βοηθητικό ε, για να δει κανείς σε ποιο βαθμό οι γενικές αρχές και αξίες διακυβεύονται ή όχι. Ο νόμος αυτός κάποιες, ο αυτός προβλέπει κάποιες εγγυήσει για τη διαφύλαξη αυτών των αρχών και των αξιών και φορώντας πάντα το ουγγαρέζικο καπέλο μου σας λέω ότι εμείς δίνουμε αυτές τις εγγύησεις ώστε να είναι απολύτως ξεκάθαρη η κατάσταση. Παρά τις παρεξηγήσεις, παρά τις διαστρεβλώσεις και τον πολύ ζωηρό, θερμό πολιτικό διάλογο, ε, διάλογο εξαιτίας αυτού του θέματος. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα τώρα. Ε, πρέπει να σας παραπέμψω στα όσα είπα, ε, είπα για το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ της είπα της εκπροσώπου και του Συμβουλίου και του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Όσον αφορά στο εμπάργκο, είναι κάτι που αφορά τις χώρες μέλη. Οι χώρες μέλη το συζητούν από καιρού καιρών και οι χώρες μέλη μέχρι τώρα έχουν καταλήξει σε μια κοινή θέση στο ίδιο κοινό συμπέρασμα που ισχύει και που αποτελεί την ε, ισχύουσα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισλανδία. Ποια κεφάλαια θα ανοίξουν. Συνήθως αρχίζουμε με τα πιο απλά κεφάλαια και μετά προχωράμε στα πιο δύσκολα. Η Ισλανδία όμως είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, διότι ε, δεν θέλω βέβαια να προβλέψω τίποτα, σας παρακαλώ μην ομένω αυτά που λέω, αλλά κάποια κεφάλαια ίσως ανοίξουν και κλείσουν ταυτόχρονα, διότι σε τελευταία ανάλυση τα ε, ε, κριτήρια έχουν εκπληρωθεί τα κριτήρια έχουν εκπληρωθεί, οι στοχοδείκτες έχουν τεθεί. Ίσως λοιπόν συμβεί κάτι τέτοιο και να μπορεί να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις τα πιο δύσκολα κεφάλαια που περιλαμβάνουν ε, πιο λεπτά και ευαίσθητα ζητήματα. Σερβία, Κωσυφοπέδιο, συνομιλίες. Προτρένουμε, προτρέπουμε αμφότερες τις πλευρές και η ύπατη εκπρόσωπος έλαβε αρκετά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ότι οι συνομιλίες πρέπει να αρχίσουν το ταχύτερο δυνατό. Ε, και εγώ διατύπωσα προσωπικά διατύπωσα μια λύπη, τη λύπη μου, ότι οι συνομιλίες αυτές δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει. Δεν θέλω να επιρρύψω την ευθύνη σε καμία πλευρά. Πάντως το ότι δεν ξεκίνησαν οι συνομιλίες είναι γεγονός. Πάντως εμείς ε, προτρέπουμε αμφότερες τις πλευρές ότι πρέπει να ξεκινήσουν οι συνομιλίες με τα ευκολότερα, τα πιο τεχνικής φύσεως ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με το ζήτημα του καθεστώτος, που όμως θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που ζουν εκεί και που ζουν όλα τα προβλήματα επικοινωνίας, βασικής στοιχειώδους ασφάλειας κλπ. Πρόθεσή μας λοιπόν είναι να ενθαρρύνουμε τα μέρη να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις το ταχύτερο. Το ταχύτερο δυνατό. Τουρκία. Αναφέρθηκε από διάφορους συναδέλφους. Υπάρχουν τρία κεφάλαια, θεωρητικά, που θα μπορούσαν να ανοίξουν. Ενέργεια, ε, κρατικές προμήθειες και κοινωνικά ζητήματα. Όλα θα μπορούσαν να ανοίξουν ή οποιοδήποτε από αυτά θα μπορούσε να ανοίξει, αλλά προφανώς υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, κάποιες δυσκολίες με τα κριτήρια. ε μπορώ λοιπόν να υποσχεθώ ότι οποιοδήποτε από τα τρία αυτά θα μπορούσε να ανοίξει. Αυτό όμως που μπορώ να υποσχεθώ και δεσμεύομαι γι' αυτό είναι ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τουλάχιστον, τουλάχιστον να μπορέσουν να ανοίξουν τα κεφάλαια. Πρέπει να τελειώσω, αντιλαμβάνομαι, αλλά μια τελευταία λέξη. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Λάσλο Τάρκης που αναφέρθηκε στο θέμα της στρατηγικής του Δούναβη, διότι είναι το καλύτερο σύμβολο, η καλύτερη επίδειξη της συμπεριληπτικής φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει να κάνει μόνο με την διεύρυνση, είναι μια μακροπεριφερειακή στρατηγική που περιλαμβάνει πολλές περιφέρειες, 14 χώρες, 8 εκ των οποίων είναι μέλη και 6 που δεν είναι μέλη. Αυτό αφεαυτού είναι ένα μήνυμα που δείχνει ότι δεν θέλουμε να ανεγείρουμε ένα, ένα τείχος μεταξύ μελών και μελών. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό και σύμβολο ε, πολύ επιτυχούς περιφερειακής συνεργασίας. Δεν έχω χρόνο να αναφερθώ στην πολιτική ανατολικής γειτονίας. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι ότι υπόσχομαι να ξανάρθω, θα ξανάρθω και προσβλέπω στις ερωτήσεις σας και στις ε, αυστηρές σας επικρίσεις και κριτικές που δεν τις είχα αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις καλές ευχές σας και θα ήθελα για μία ακόμα φορά να εκφράσω την επιθυμία μου να συνεργαστούμε ε, στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Λίγη η συζήτησή μας με την κοινή αυτή ευχή να μπορέσουμε να αναπτύξουμε θέματα που είναι δική σας αρμοδιότητας Χαιρόμαστε που σας γνωρίσαμε εκ του σύνεγγης. Είσαστε άκρος συμφιλιωτικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή εργασία για το επόμενο εξάμεινο. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Θα διακόψουμε για λίγα λεπτά. Colleague, please uh, sit down. We have to start because uh, uh, Κυρίες και έχει έρθει ο Επίτροπος και δεν έχουμε και πολύ χρόνο να συζητήσουμε μαζί του. Θα ήθελα λοιπόν να τον καλωσορίσω, να καλωσορίσω τον φίλο μας, τον έλεγα πλέον, γιατί εδώ και αρκετό καιρό έρχεται να μας επισκεφτεί με πνεύμα συνεργασίας και οι ε, βουλευτές από την Αρμενία, τη Γεωργία, την ε, ε, Μολδαβία βρίσκονται εδώ στην αίθουσα και τους καλωσορίζουμε. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για την πολιτική γειτονίας. Αυτό είναι το θέμα που θα εξετάσουμε σήμερα και το εξετάζουμε το θέμα με τον αρμόδιο, τον καθήλυνα αρμόδιο. ξεκινάμε όμως με κάτι πολύ ενδιαφέρον και θα ακούσουμε την ομιλία του βέβαια, να το πω αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα να πούμε σε εσά, κύριε Επίτροπε, κάποιες ε, θέσεις ε, των ε, Ευρωβουλευτών Νταβίτ και Σίβιτσικ που έχουν επεξεργαστεί προτάσεις ψηφίσματος ως εισηγητές και θα τις παρουσιάσουν αυτές κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες. Άρα δηλαδή αν θέλετε πρόκειται για ένα είδο διμερούς ανταλλαγής απόψεων για θέματα που αφορούν τις δικές σας τις απόψεις και αρμοδιότητες, αλλά και τις δικές μας. Στις 26 ε, Οκτωβρίου μας ε, παρουσιάσατε τις ε, φάσεις, τα βασικά σημεία για την εξέλιξη της πολιτικής γειτονίας και σήμερα λοιπόν έχουμε περαιτέρω εμβάθυνση του θέματος. Δεν θα ήθελα να σας καθυστερήσω περαιτέρω στην παρέμβασή σας. Θα ήθελα να είσαστε όσο πιο περιεκτικός γίνεται για να μπορέσουμε όλοι μας, κυρίως οι συγητές τους οποίους προανέφερα, να ε, αναπτύξουν με σας ε, διάλογο και να συνεργαστείτε. Σε εσά κύριε Επιτροπεολόγος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη και αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, για μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Στις 26 Οκτωβρίου Ήδη τότε ανταλλάξαμε απόψεις ε, για θέματα που προκύπτουν από την αναθεώρηση. Πριν λοιπόν ακούσω τις δικές σας απόψεις, ε, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω σύντομα ε, τις κατά την άποψή μας βασικές ερωτήσεις, τα βασικά θέματα που προκύπτουν μέχρι σήμερα από την αναθεώρηση. Μέχρι τώρα λοιπόν βάλαμε τρία ερωτήματα στους εταίρους μας σε κράτη-μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Πρώτα, το μακροχρόνιο όραμα της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Δεύτερον, πιο συγκεκριμένοι στόχοι σε διάφορους τομείς, ε, μεσοπρόθεσμα. Και τρίτον, τα εργαλεία και οι πόροι που χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ περαιτέρω στα θέματα αυτά. Όσον αφορά τη μακροχρόνια αναθεώρηση, υπάρχει κοινό όραμα με τους γείτονές μας. Χώρος, πολιτική συνεργασία και οικονομική ολοκλήρωση. Όσο πιο μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση γίνεται. Οι εταίροι μας βεβαίως υπογράμμισαν το ότι είναι απαραίτητο ε, να ε, προκύψουν περισσότερα ωφέλη και στήσαν την προσοχή τους σε δεσμεύσεις ε, για μεταρρυθμίσεις. Όλοι δεσμεύτηκαν για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και για, την, για το κράτος δικαίου. Αυτά πρέπει να είναι σημαντικά στοιχεία, καθοριστικά στοιχεία της πολιτικής. Είτε δούμε προς Ανατολάς είτε προς Νότον υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που δείχνουν ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να στηρίξουμε τις φιλοδοξίες των εταίρων ε, και φίλων μας. Μία πρόταση είναι ε, το μακροχρόνιο μοντέλο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας θα πρέπει να είναι ο ευρωπαϊκός οικονομικός χώρος. Αυτό ε, είναι ε, μία πολύ φιλόδοξη δομή ένα μόρφωμα το οποίο απαιτεί από τους εταίρους να δεχτούν κάποιους ε, περιορισμούς ε, στις, ε, στις αποφάσεις που λαμβάνουν. Και από πολιτική και οικονομική πλευρά αυτό είναι εφικτό για τους εταίρους μας. Ένα άλλο θέμα είναι πώς η μακροχρόνιες οικονομικές στρατηγικές των εταίρων μπορούν να συνδυαστούν καλύτερα με τις δικές μας. Αυτό είναι κάτι επί του οποίου θα είναι πολύ χρήσιμες οι απόψεις σας. Και τέλος, οποτεδήποτε γίνεται λόγος για περισσότερο φιλόδοξες προσφορές, αναπόφευκτα καταλήγουμε στο θέμα της ε, διαφοροποίησης. Οι περισσότερες ε, εκθέσεις ε, επιμένουν στο θέμα αυτό και συμμερίζομαι απόλυτα αυτό που είπε ο κύριος Σίβιετς στην έκθεσή του για το πώς μπορεί κανείς να ενισχύσει τους δεσμούς ε, με τους ε, βέλτιστα αποδίδοντες εταίρους και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τους άλλους. Μπορούμε να είμαστε πιο αυστηροί στον τρόπο που εφαρμόζουμε τη διαφοροποίηση και Πώς πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να γίνει στην πράξη. Αν πάμε σε πιο συγκεκριμένους ε, μεσοπρόθεσμους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, ε, χαιρετίζω την δική σας ε, τη συνεισφορά σε τέσσερα θέματα, κυρίως στη διακυβέρνηση, στις προστατευόμενες συγκρούσεις, οικονομική ολοκλήρωση και κινητικότητα. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, Πώς μπορούμε λοιπόν να ενισχύσουμε το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα έτσι ώστε να προάγουμε τη συμβατότητα με τους στόχους, της Προδιαγραφής του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δικαστική εξουσία για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τη διαφθορά και πώς μπορούμε να ε, ε, ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών, όπως πολύ σωστά αναφέρεται και στην ε, έκθεση. Οι εταίροι μας ε, ζητούν από μας να αναβαθμίσει τις δράσεις της. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα νέα εργαλεία της συνθήκης της Λισαβόνας για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Όσον αφορά την οικονομική ολοκλήρωση, η ενσωμάτωση καθυστερημένων περιοχών είναι στόχος ε, για τους εταίρους μας και προς Ανατολάς και προς Νότον. Ε, αυτό το εργαλείο πρέπει να προσαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να καλύπτει τις ε, ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ε, ε, εταίρων μας. Όσον αφορά την κινητικότητα, πρέπει να δούμε τις παραμέτρους που μπορούν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου όλοι θα κερδίζουν από την κινητικότητα και την ασφάλεια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες και τα αιτήματα των εταίρων. Ποιε είναι οι προϋποθέσεις για την πρόοδο στην κατάργηση προξενικών θεωρήσεων υπάρχει χώρος για πιο πρακτικές προτάσεις ε, όσον αφορά την ε, κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Και τέλος, όσον αφορά τους πόρους, είναι απαραίτητο τους στόχους μας να τους μετατρέψουμε σε πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για πολλά κράτη-μέλη. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν επαρκή χρηματοδότηση κατά την επόμενη δημοσιονομική προοπτική για να ε, καλύψουμε ε, τους στόχους της ε, πολιτικής μας. Και χαίρομαι που όλοι απαιτούν να υπάρχει αυτή η σωστή χρηματοδότηση. Για να γίνει αυτό προφανώς χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας και πάλι λοιπόν η ιδέα σας είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες όχι μόνο για τη χρηματοδότηση αλλά και για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την παροχή της βοήθειάς μας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι για την Υπουργική Διάσκεψη που ε, προγραμματίζουμε για την επόμενη εβδομάδα. Από την εμπειρία σας γνωρίζετε ότι το να συγκεντρώσει κανείς όλους τους Υπουργούς Εξωτερικών της περιοχής δεν είναι εύκολο. Σχεδόν ε, όλοι οι οι ομόλογοι μας μας είπαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν μπορούν να έρθουν γιατί πρέπει να πάνε ε, στην ε, συνάντηση στο Κατάρ με θέμα την Ιερουσαλήμ. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι δεν ήταν κατάλληλη χρονική στιγμή και αποφασίσαμε να ε, αναβάλουμε αυτή τη συνάντηση. Αυτό βέβαια δεν μας εμποδίζει στο να συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Στις 20 Απριλίου πρέπει βέβαια να δημοσιεύσουμε την ανακοίνωσή μας. Αυτά προς το παρόν είχα να σας πω. Τώρα πρέπει να σας ακούσω. Ξέρω ότι έχετε ορίσει δύο συγητές και γνωρίζω ότι οι δύο αυτοί οι έχουν ήδη ολοκληρώσει το έργο τους. Με χαρά να ανταλλάξουμε σήμερα απόψεις, τις πρώτες απόψεις και θα αποδώσω ιδιαίτερη σημασία ε, στις, ε, στα μελλοντικά σας ε, ψηφίσματα. Ελπίζω λοιπόν η σημερινή συζήτηση μαζί με όλα τα άλλα που έχουν προηγηθεί να μας προσφέρει ικανοποιητική τροφή για σκέψη έτσι ώστε να προάγουμε τις φιλόδοξες προτάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Όπως ε, είπαμε στην αρχή της συνάντησης, σήμερα δεν έχουμε μόνο να ακούσουμε, αλλά και να προτείνουμε κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σίβιτς. Θα ήθελα να αρκεστείτε στα πέντε λεπτά έτσι ώστε να γίνει η ευρύτερη δυνατή συζήτηση. Κύριε Σέβιτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Επίτροπε για αυτή την παρουσίαση. Έχει μεγάλη σημασία το πώς παρουσιάζεται το θέμα. Το παρουσιάσατε πολύ καλά ε, διαρθρωμένο. Νομίζω ότι μέχρι τούδε φτάσαμε σε πολύ καλά αποτελέσματα και στο σχέδιο έκθεσης ακολουθήσαμε τις τρεις ερωτήσεις που ετέθησαν και σήμερα. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ εισηγητής μαζί με τους σκιώδεις από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Το, το έργο μας έχει κάπως διευκολυνθεί. Έχουμε αρκετά διευκολυνθεί και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ότι η πολιτική γειτονίας που πρώτο προτάθηκε το 2004 αφορούσε τη μεγάλη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως πολλοί βρέθηκαν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν προσχώρησαν, αλλά βρέθηκαν πολύ κοντά. Μέσα στα 7 χρόνια που ακολούθησαν η κατάσταση άλλαξε δραματικά και η πολιτική γειτονία κατέδειξε ότι αλλάζουν και οι ανάγκες των εταίρων μας. Θα ήθελα να τονίσω ότι κατά τα 7 αυτά χρόνια σε σχέση με τους ε, προσανατολάς εταίρους είδαμε πολλές δραματικές αλλαγές, θετικές βεβαίως, όπως η ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ουκρανία, αλλά και αρνητικές τάσεις όπως είδαμε στην περίπτωση της Λευκορωσίας. Άρα δεν κινούνται όλα προς ε, τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν ε, πολλά σκαμπανεβάσματα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι στη Βόρειο Αφρική σήμερα, στις χώρες Μαγκρέμπ, πέφτει το τείχος, διότι υπήρχε ένα τείχος προστασίας των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει κατατροποθεί, ιδιαίτερα στην ε, Ισία. Άρα τα επόμενα πέντε χρόνια θα πρέπει να δράσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, στις προκλήσεις στην Ουκρανία, στη Μολδαβία και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Φέρουμε μεγάλη ευθύνη, διότι θα πρέπει να είμαστε θαραλέοι και υπεύθυνοι. Και το ε, μήνυμα που θα αποστείλουμε θα πρέπει να είναι θετικό όχι μόνο για τους κυβερνήτες αλλά και για τα έθνη. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα τα σημεία του σχεδίου έκθεσης. Θα ήθελα να πω ότι θα θέλαμε να συνεχιστεί η πολιτική γειτονίας. Είναι μια πολιτική που αφορά και τις εταιρικές σχέσεις προς Ανατολάς θα θέλαμε να γίνει μια έξυπνη διαφοροποίηση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή πολιτική προς Ανατολάς και προς Νότον, διότι τα προβλήματα είναι παρόμοια. Μιλάμε για ανθρωπινά δικαιώματα, για δημοκρατία, για βασικές ελευθερίες. Οι κοινωνίες είναι διαφορετικές, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν οι ίδιες. Αν ε, αναζητήσουμε κάτι καινούριο στην έκθεση σε σχέση με την κατάσταση λίγο χρόνια πριν, το μόνο καινοτόμο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε άμεση επαφή με την κοινωνία, με τους νέους, με τα μέσα επικοινωνίας, να έρθουμε σε επαφή με την, τις τοπικές κυβερνήσεις σε μια γλώσσα που να είναι κατανοητή από τους ανθρώπους. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε την κυβέρνηση συγκεντρωτικά, σε κεντρικό μόνο επίπεδο. Θα θέλαμε να διευκολύνουμε αυτές τις τάσεις και τις υποδομές. Διαφορετικά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Θα πρέπει να άρουμε αυτά τα προσκόμματα έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις επιμέρους κοινωνίες. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο ανέφερε ο Επίτροπος, το θέμα της χρηματοδότησης. Εμείς θα πρέπει να αναφερθούμε στο τι ποσά είμαστε έτοιμοι να δαπανίσουμε. Βέβαια, η καιρή είναι δύσκολη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να δαπανηθούν κονδύλια. Και ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι το εξής. Θα πρέπει να δούμε ποιες ε, είναι οι προσδοκίες αυτών των κρατών, των υποψηφίων κρατών. Και αυτό δεν μπορούμε να τους το αφαιρέσουμε εάν δεν προσφέρουμε κάτι το συγκεκριμένο ως προς την ένταξή τους, τότε δεν θα μπορέσουμε να τις διευκολύνουμε αν δεν υπάρχει αυτή η προοπτική. Και ως προς τα τελικά μου σχόλια, θα ήθελα να πω ότι Μέσα στα πλαίσια της Euronest θεωρήσαμε ότι και η Euronest θα πρέπει να είναι ένας εταίρος. Πρόκειται για το κοινοβουλευτικό αυτό σκέλος, το οποίο θα θέλαμε να προωθήσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές με τους οποίους ήρθα σε επαφή, καθώς και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που με βοήθησαν ιδιαίτερα ως προς τη συνεργασία επί αυτού του θέματος. Αυτό που προβάλλουμε σήμερα είναι ένα προσχέδιο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη εντολή, αλλά νομίζω ότι θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα και θα βοηθήσει και τον ε, Επίτροπο. Ευχαριστούμε κυρία Σίβιτς. Το λόγο έχει ο κύριος Σαλαφράνκα, ο οποίος θα μας μιλήσει εξ ονόματος του κυρίου Ντέιβιντ σε σχέση με την μεσογειακή διάσταση, διότι ο υπεύθυνο δεν είναι εδώ και θα μας μιλήσει εξ ονόματος του ΕΛΚ και ιδιαίτερα με, ως προς την έκθεση Σίβιτς για την ανατολική διάσταση. Θα Είμαι ιδιαίτερα σύντομος, διότι ο κύριος ε, Ντέιβιντ είναι άρρωστος και δεν μπορούσε να έρθει εδώ. Και γι' αυτό μου ζήτησε να παρουσιάσω μου ζήτησε να παρουσιάσω τις θέσεις του και επίσης η κυρία Γιαννάκου μου ζήτησε να την εκπροσωπήσω γιατί βρίσκεται σε μια άλλη επιτροπή. Θα ήθελα εξ ονόματος των δύο αυτών μελών, των δύο μελών και της πολιτικής μου ομάδας να καλωσορίσουμε καταρχήν τον κύριο Φούλε. Ε, χαιρόμαστε διότι είχε επαθές με τα μέλη του Κοινοβουλίου καθώς και τα Εθνικά Κοινοβούλιο και εκπροσώπους τρίτων χωρών. Οι δύο εισηγητές και οι ισχυώδεις συνεργάστηκαν έτσι ώστε να δώσουμε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για να καλύψουμε τις δύο αυτές γεωγραφικές ζώνες. Καταρχήν, θεωρούν ότι θα πρέπει να εντάξουμε συγκεκριμένους στόχους στην πολιτική γειτονίας, δηλαδή να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους και να λάβουμε υπόψη το γράμμα των συνθήκων έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις αξίες που μας διέπουν. Ο κύριος ε, Ντέιβιτ και η κυρία Γιαννάκου ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις γείτονες χώρες καθώς και μια περιφερειακή συνεργασία. Επειδή μιλάμε για τη ε, νότια διάσταση της πολιτικής ε, γειτονίας, ο κύριος Ντέιβιτ ανέφερε ότι θα πρέπει να τονίσουμε το θέμα της Ένωσης για τη Μεσόγειο και, και εκφράζει τη λύπη του διότι δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί η δεύτερη διάσκεψη όπως θα θέλαμε. Επίσης ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να εντάξουμε την Ένωση για τη Μεσόγειο σε μια συνολική στρατηγική. Και υποστηρίζει τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τη δίωξη των χριστιανών. Θεώρησε λοιπόν ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να, να προωθηθεί και να στυλιτευτεί κατάλληλα. Ως προς την, την Ισία, δεν αναφέρθηκε ειδικά σε αυτήν, διότι ε, το θέμα παραμένει σχετικά παρχαιωμένο με βάση τα νέα δεδομένα. Είχαμε συναντήσεις με τους σκιώδεις και σε σχέση με το τμήμα της κυρίας Γιαννάκου, με το θέμα της κυρίας Γιαννάκου υπάρχουν δύο σχόλια ειδικά ως προς την παράγραφο 18, όπου αναφέρεται ότι η αύξηση των κονδυλίων αποτελούν ένα μέσον και μηχανισμό για να προωθήσουμε αυτά τα μέτρα. Η κυρία Γιαννάκου θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν όροι και ένας κανόνας αιρεσιμότητας σε σχέση με τον δημοσιονομικό έλεγχο για να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτά τα μέσα και τους πόρους προς τις γείτονες χώρες. Ως προς την προσανατολάς διάσταση, η πολιτική γειτονίας θα προβάλλει λύσεις στις σειράξεις που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή και μέσω ΟΑΣΕ και μέσω άτυπων επαφών στις γείτονες αυτές χώρες, εκεί ιδιαίτερα που υπάρχουν σειράξεις και κλειδονισμοί, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε ένα νέο μέσο γειτονίας και να χρησιμοποιήσουμε και τις καλές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Θα ήθελα να επαναλάβω εξ ονόματος των ε, δύο μελών του ΕΛΚ ότι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί σας για να λάβουμε υπόψη κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνεργασία αυτή προς Νότον και προς Ανατολάς. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαλαφράγκα. Το λόγο έχει ο κύριος Πάσκου για δύο λεπτά. Ο αντιπρόεδρος ο κύριος Πάσκου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να επισημάνω το γεγονός ότι είστε διαθέσιμος και η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και ημών, κυρία Επίτροπε, είναι υποδειγματική και ελπίζουμε ότι δεν θα μεταβληθεί στο μέλλον. Ελπίζουμε να μπορούμε να σας εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά πιο συχνά. Στην περίπτωση της Τινησίας, δια... ανακαλύψαμε ότι ο λαός θεωρούσε αυτό το καθεστώς διεφθαρμένο και το εξεδίωξε, το ξεφορτώθηκε. Αλλά από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είχαμε ακούσει τίποτα σε αυτό το κοινοβούλιο. Και τώρα διαβάζουμε στο τύπο ότι έχουν διαρρεύσει έγγραφα από πλευράς, ε, έγγραφα που έχουν να κάνουν με την Παλαιστινιακή Αρχή και ε, υπάρχουν ε, κατηγορίες ότι γίνεται διασπάθηση χρημάτων κλπ. Και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να φτάσουμε μια μέρα εμπλεκόμενοι και εκεί. Ξέρουμε όμως ότι οι διαπραγματεύσεις επί του Μεσανατολικού έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Πώς τώρα εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάνουμε κάτι ώστε να άρουμε αυτό το αδιέξοδο. Τι κάνουμε. Και η συνθήκη η οποία ακόμα κρεμεί. Αν προχωρήσει θα είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο για να διαδραματίσουμε έναν πιο επικοδομητικό ρόλο. Η κυρία Μπραντνερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Uh, just two points I want to mention. One, you were asking about Επειδή μιλήσατε για την κοινωνία των πολιτών και την στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία. Ε, ασφαλώς χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για την υποστήριξη της κοινωνίας των ε, πολιτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της ενδιαφερόμενης κυβέρνησης και στην Αφρική αυτό χρειαζόμαστε και νομίζω ότι θα συζητήσουμε το θέμα της Τινησίας αργότερα, αλλά πρέπει να ζητήσουμε ε, κονδύλια ώστε να κάνουμε περισσότερα και ίσως μειώσουμε τα κονδύλια σε άλλα θέματα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Δεν μπορούμε διαρκώ να ζητάμε περισσότερα χρήματα, αλλά πρέπει να θέσουμε ε, προτεραιότητες και να λειτουργήσουμε με βάση αυτέ. Η στρατηγική λοιπόν δεν είναι να ζητάμε περισσότερα, αλλά να θέτουμε προτεραιότητε και ε, διότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρξουν περικοπές. Ε, ε, και δεν θα πρέπει να ε, επιδιώκουμε άμεση ενίσχυση του προϋπολογισμού, όπως ας πούμε σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Αφρικής. Ε, πρέπει να στηρίζουμε περισσότερο ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις κλπ. Πρέπει να χρηματοδοτούμε οργανισμούς οι οποίοι ελέγχουν το τι γίνεται με τα δικά μας λεφτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μπραντνα. Τζάλα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ε, με βάση την έκθεση του κυρίου Μαρατσίνη θα ήθελα να ε, θέσω το ερώτημα στον Επίτροπο. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ εμπεριστατωμένο σχέδιο κειμένου και έχω απλώς δύο σύντομα σχόλια. Πρώτον, Συμφωνώ απολύτω με τον εισηγητή ότι πρέπει να γίνει σαφή διαφοροποίηση με επί τη βάση της προόδου των χωρών. Συνεπώς, αυτοί που έχουν καλύτερες επιδόσεις να έχουν πιο απτή στήριξη στον τομέα ε, του εμπορίου, της θεωρήση διαβατηρίων ή τον πολιτικό διάλογο και στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι είναι χρήσιμο να αναφέρουμε με σαφήνεια πώς θα πάει η Μολδαβία διότι η Μολδαβία είναι μια πετυχημένη ιστορία, ε, ιδιαίτερα πέρσι, και πρέπει να την επιβραβεύσουμε. Δεύτερον, για μένα είναι πρόβλημα που η έκθεση δεν αναφέρει καθόλου τη Ρωσία. Αντιλαμβάνομαι ότι η Ρωσία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων στην ανατολική γειτονία, στην πολιτική γειτονία, στην ανατολική της διάσταση. Ευθύ εξ αρχή η Μόσχα εξέφρασε σκεπτικισμό και άσκησε κριτική ε, ως προς την πολιτική γειτονία. Αλλά σταδιακά η στάση της Ρωσίας άλλαξε. Και η Ρωσία ε, συμμετέχει σε μια άτυπη ομάδα των φίλων της Ανατολικής Γειτονίας. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε χρήση αυτής της ευκαιρίας και να ενθαρρύνουμε την Ρωσία να συμμετάσχει στις δραστηριότητες της Ανατολικής Γειτονίας και στα προγράμματα. Η αυξημένη συμμετοχή της Ρωσίας όχι μόνο θα ενισχύσει την αξιοπιστία της πολιτικής γειτονίας προς Ανατολάς, αλλά θα έχει και θετικές συνέπειες στις διμερείς μας σχέσεις με την Ρωσία. Νομίζω ότι αξίζει η Ρωσία ε, μίας μνήας στην έκθεση αυτή και είναι μια υπενθύμηση και προς τον Επίτροπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστούμε τον κύριο Μπάλα. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Τάνακ ε, γιατί έπρεπε να του δώσω προηγουμένως ε, ε, το λόγο και ήμουνα κάπως αφηρημένος. Και εγώ είμαι σκιώδης. Ήμουν δύο φορέ εισηγητή σχετικά με την πολιτική γειτονία στο προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Στην αρχή υπήρχε ένα εισηγητής για ολόκληρη την πολιτική γειτονία και στη συνέχεια δύο συνπροέδρους για την ανατολική διάσταση και την νότια. Και τώρα έχουμε δύο ξεχωριστέ εκθέσει. Αυτό δείχνει και είναι προβλέψιμο ότι όλο και περισσότερο το Κοινοβούλιο και οι Κομισιόν ε, δίνουν ιδιαίτερη σημασία διότι το, το Μαρόκο και η Ορδανία και οι άλλες χώρες έχουν αυξημένο ενδιαφέρον. Βεβαίως τώρα έχει μία σχέση, ε, μάλλον κοινά σύνορα ή όμορα σύνορα. Ε, και το Καζακστάν ενδεχομένως θα μπορούσε να περιληφθεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν αλλάξει πορά από το 2006 όταν άρχισαν να εξετάζουν αυτή την πολιτική. Η ε, Ουκρανία δεν είναι καν μία ενδυνάμει υποψήφια χώρα, ε, ενώ η Αλβανία είναι, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι σκοτώνται στους δρόμους, ούτε η Μολδαβία επίσης και ως προς την ε, Ουκρανία κάτω από την κυβέρνηση του Κόβετς φοβούμε ότι δεν μοιραζόμαστε κοινέ αξίες. Όλες οι παγωμένες διενέξεις παραμένουν παγωμένες εκτός ενδεχομένως από τον Ακόρνο Καραμπάχ και το ε, Αζερβαϊτζάν που το Αζερβαϊτζάν όλο και πιο ε, ε, αισθάνεται όλο και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και η Γεωργία η οποία είναι οικονομικά η πιο προχωρημένη, η πιο διαφανής και με τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις αυτή τη στιγμή είναι υπό ρωσική κατοχή. Στο Νότο χριστιανοί διώκονται σε χώρες όπως η Αίγυπτος, αλλά ακόμα και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Είμαι εξαιρετικά λοιπόν ε, απογοητευμένος σχετικά με την πολιτική, αλλά σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας. La parola all'onorevole πρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας για τη σχέση με τη Λευκορωσία. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αρχίσω με τα συγχαρητήρια προς όσους συντάσσουν τις δύο εκθέσεις, ιδιαίτερα στον Πολωνό συνάδελφο, παρά το γεγονός ότι ανήκω σε διαφορετική πολιτική παράταξη. Ε, η έκθεση του κυρίου Σίβιετ για την ανατολική διάσταση της πολιτικής γειτονίας ε, βρίσκεται πολύ κοντά στα δικά μου ενδιαφέροντα. Ιδιαίτερως θα ήθελα να, συγχα... να τον συγχαρώ για το γεγονός ότι επισημαίνει τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών στην έκθεση. Και τονίζει σε μία από τις παραγράφους ότι θα πρέπει Θα πρέπει η ευρωπαϊκή πολιτική με τρόπο ενεργό να εφαρμόσει την πολιτική της προς Ανατολάς. Τώρα, σχετικά με τα θέματα που έθεσε ο Επίτροπος ως προς το όραμα και το θέμα που έθεσε ο κύριος Σιβίτς για την συμμετοχή. Συχνά μας κατηγορούν ότι χρησιμοποιούμε διπλά standards έναντι των γειτόνων από Ανατολάς προς Νότον. Κάποιους τους μεταχειριζόμαστε ως Ευρωπαίους γείτονες, και άλλους όχι. Ε, πρέπει λοιπόν η προοπτική της ε, συμμετοχής ε, να αποτελέσει κίνητρο για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποστινάου ε, που είναι εισηγητής για την Αλβανία και την επόμενη φορά έχουμε προβλέψει εδώ στην ΑΦΕΤ ακριβώς μια συζήτηση για την κατάσταση στην Αλβανία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, η δική μου ερώτηση δεν αφορά την ε, ε, Ανατολική Γειτονία αλλά την Αλβανία γιατί ε, το θέμα είναι φλέγον και εσείς ξέρετε καλύτερα από όλους τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα πέρυσι. Την Παρασκευή επιτέλους ξεκίνησε ο διάλογος αλλά με σφαίρες στα, τύρανα και αυτό πρέπει να ανησυχεί όλους Εδώ λοιπόν και αρκετούς μήνες εσείς προσπαθείτε να διευκολύνετε το διάλογο ανάμεσα στα δύο μέρη, να αναζητηθεί μια λύση ε, στο αδιέξοδο που υπάρχει στα τυραννά εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Είχατε επίσης επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον με τις δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες, το ΕΛΚΑ και τους ε, σοσιαλιστές. Όμως τελικά δεν επιτέχθηκε καθόλου πρόοδος. Γι' αυτό λοιπόν, όσο έχει σήμερα η κατάσταση στην Αλβανία, εσείς πώς την αξιολογείτε και δεύτερον, τι πρέπει να γίνει για να αποτραπεί η ε, το εκρηκτικό τέλος της κατάστασης και τελικά, τελευταία ερώτηση, αν δεν υπάρξει λύση, τι θα κάνουμε. Ευχαριστούμε. Βάγγελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές ε, και όσους μίλησαν στη σημερινή συζήτηση, αλλά θα ήθελα και εγώ να είμαι σύντομος λέγοντας το εξής, ότι η νότια διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας επισκιάζεται αναμφίβολα από τα ανεπίλητα προβλήματα της περιοχής. Μιλάμε για την Μεσογειακή Ένωση, η οποία όμως ε, δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει. και οποτεδήποτε γίνονται συζητήσεις ε, υπό την αιγίδα της Μεσογειακής Ένωσης εμπλεκόμεθα σε αυτές τις ε, συζητήσεις για τη Μέση Ανατολή και όλοι γνωρίζουν ότι δεν οδηγούν πουθενά. Κύριε Επίτροπε, αυτά τα θαυμάσια έγγραφα. Εξαρτώνται βέβαια από το κατά πόσον θα μπορέσουμε να λύσουμε κάποια προβλήματα. Γιατί αλλιώς τέτοιου είδους ε, πρωτοβουλίες δεν μπορούν να τελεσφορήσουν. Σήμερα πήρα ένα μήνυμα ότι ο Γενικός Γραμματέας της ε, Ένωσης για τη Μεσόγειο παρετήθηκε Και είχα ε, εκπλαγεί και όταν δέχτηκε τη θέση, ήταν 42 χρονών. Αυτή είναι μια θέση για κάποιους σαν και εμένα που ε, σύντομα πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Δεν εξηγεί γιατί ε, αποσύρθηκε, αλλά παρετήθηκε δηλαδή, αλλά καταλαβαίνω την απογοητευσή του. Αυτή η οργάνωση έχει παραλύσει. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτά που είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι. Δηλαδή, τελικά, αν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο να λύσουμε τα φλέγοντα ε, προβλήματα της περιοχής και κάθε μέρα προστίθενται και καινούρια, τότε όλα αυτά τα προγράμματα καταρτίζονται και συζητιούνται επί Ματέο. Σούλτς, δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για το ότι ε, έχετε στενές επαφές με την Επιτροπή μας. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουμε επίκαιρες ερωτήσεις. Ήσασταν παρόν και στην έκτακτη συνάντησή μας ε, όταν ε, η, έγινε η έκθεση της ε, Λευκορωσίας και πολύ συχνά πολλοί ζητάνε να ανασταλούν οι σχέσεις με τη χώρα αυτή. Εσείς πώς αξιολογείτε τις σχέσεις με τη Λευκορωσία, τελικά τι καταφέραμε και η αναστολή είναι εργαλείο για να ασκείται πολιτική πίεση. Και ένα άλλο ερώτημα. Ε, τον κύριο Φαν Ρόμπεϊ τον ρώτησα κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο όπως η δυτικοεφρανική ένιση η οποία ε, πήγε στην ακτή του ελεφαντοστού για να τους ε, βοηθήσει, για να δει τι γίνεται. Μήπως θα έπρεπε και ο κύριος ε, Μπαρόζο ε, και η κυρία Άστον να πάνε στον Λουκασέγκο για να του εκφράσουν με σαφήνεια την άποψή τους. Είπε ότι η συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη ενδείκνυται για να ε, λογοδοτήσει ο Λουκασέγκο. Μόνο που ο Λουκασέγκο δεν δικαιούται να πάει στη Βουδαπέστη και το ίδιο συνέβη και στην Πράγα το 2009 όταν δεν μπόρεσε να πάει για να συμμετάσχει στην συνάντηση για την ε, πολιτική γειτονία. Εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι στη Βουδαπέστη ε, πρέπει να έρθει ο Λουκασέγκο να του ζητηθεί ο λόγος για όλα αυτά που έγιναν σε εκλογές και ε, όλα αυτά που ακολούθησαν. Δηλαδή πριν περάσουμε σε πιο αυστηρές κυρώσεις να αναζητήσουμε τουλάχιστον έναν ειλικρινή διάλογο. Ο Μπιόλς, εισηγητής, σκιώδης εισηγητής για τις ε, σχέσεις γειτονίας με τον Νότο. Δύο λεπτά. Ε, ε, Τρία σχόλια. Καταρχήν, ε, εδώ και κάποια χρόνια στην σοσιαλιστική ομάδα επανειλημμένα επιμείναμε ότι είναι ζωτικής σημασίας η ισορροπία μεταξύ της ανατολικής διάστασης και της νότιας διάστασης της πολιτικής μας γειτονίας και ομιλώ ως σκιώδης ε, εισηγητής της έκθεσης Ντέβιτ. Χαίρομαι που υιοθετήθηκε, ωστόσο τα σχόλιά μου ξεπερνούν αυτό τα πλαίσια και θέλω να τονίσω ότι αν κανείς κοιτάξει την τρέχουσα πραγματικότητα και τα γεγονότα στη Μεσόγειο, θα διαπιστώσει ε, μια δραματική αλλαγή και τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητα στην νότια διάσταση της πολιτικής κοινωνία, όχι μόνο με τη διάθεση πόρων, αλλά επίσης ε, λαμβάνοντας μια πιο ε, ενεργητική ε, θέση πολιτικά. Ε, τα γεγονότα στην την Ισία, η ανησυχητική κατάσταση στην Αίγυπτο, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για να καταστεί σαφές ότι η κατάσταση εκεί στη Νότια Μεσόγειο είναι πάρα πολύ ασταθής για διάφορους λόγους και για διαφορετικές αιτίες υπάρχει οικονομική και κοινωνική κρίση σε όλες αυτές τις χώρες. Δεύτερο σχόλιο, πολύ σύντομο, σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην Τινησία. Η δημοκρατική επανάσταση θα πρέπει να θεωρηθεί μια ε, επιτυχημένη ιστορία ε, από εμά. Είναι πολύ σημαντικό για μας, για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ομάδα δράσης με... έτσι ώστε να υπάρξει μια πραγματική μετάβαση, δημοκρατική μετάβαση, για να παγιοποιηθεί μια πλουραλιστική δημοκρατία με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων. Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι το εξής. Ο συνάδελφος Βάγκελ το ανέφερε σήμερα μάθαμε ότι παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Θα πρέπει λοιπόν να διασαφίσουμε την κατάσταση και να δούμε ποια συνεργασία και τι τύπου συνεργασία θα μπορέσουμε να προωθήσουμε. Διακόπτει ο μιλητής. Και πώς θα δράσει η Ένωση για την Ευρώπη μαζί με τα κοινοτικά ε, όργανα, ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Νομίζω ότι αυτή η ανάγκη διαγράφεται όλο ένα και περισσότερο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι σε σχέση με την, ε, την μετά από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, ο κύριος Φίλε θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα, Άρα μπορείτε να παρέμβετε τότε για θέματα που σχετίζονται με την Τινησία. Παντζέρη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο διότι ήταν διαθέσιμο σήμερα. Μπορούμε να πούμε, για να είμαστε σαφείς, ότι η Ευρώπη έχει κλειστεί σε ένα προπύργιο, σε έναν πύργο και ε, έχει να αντιμετωπίσει και το τεστ αντοχής της διεύρυνσης και την χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό σχετίζεται και με την πολιτική γειτονία. Ξεκινώντας από αυτή τη σκέψη θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τι συμμεριζόμαστε έτσι ώστε να ξαναδούμε την πολιτική γειτονία, διότι μέχρι σήμερα ε, κατέδειξε πολλά όρια και περιορισμούς κάτι το οποίο δείχνει ότι είναι η αδύναμη εξωτερική μας πολιτική και από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε ε, κριτήρια ερεσιμότητα σε σχέση με άλλες χώρες, διότι πολλές φορές δίναμε χρήματα έναντι δημοκρατίας και αυτό είδαμε ότι δεν μπορέσαμε να το εφαρμόσουμε. Και πιστεύω ότι αυτό το μέσον θα έπρεπε να μας οδηγήσει στο να κάνουμε μία επιλογή. Δηλαδή μέσα στα πλαίσια της ε, συνεργασίας στη Μεσόγειο θα έπρεπε να βγάλουμε τη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να ορίσουμε μία ομάδα κρούσης γιατί η κατάσταση παραμένει δυσχερής και αν παραμείνει στο καζάνι της Ένωσης για τη Μεσόγειο, τότε δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Θα πρέπει να παραμείνει δηλαδή ξεχωριστό το θέμα της Μέσης Ανατολής και θα πρέπει να ορίσουμε ορισμένες προτεραιότητες, μία νέα πολιτισμική προσέγγιση. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο, και αυτό αληθεύει, μία προσωποποίηση για την ε, πολιτική οικονομικών εταιρικών σχέσεων και την πολιτική γειτονία. Βεβαίω χρειάζεται οικονομική συνεργασία, πρωτίστως περιφερειοποίηση και ούτω καθεξής. Αλλά θα πρέπει να έχουμε αυτή την προσέγγιση πρωτίστως, διότι όλα περνάνε από αυτή την κεντρική σκέψη. Ευχαριστούμε κύριε Παντσέρη. Τέλος, η κυρία Γκόμες έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο διότι βρίσκεται εδώ μαζί μας και μας απαντά. Διάβασα την εντολή διαπραγμάτευσης για την συνεργασία με τη Λιβύη και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Φαίνεται ότι το Συμβούλιο ζει σε ένα διαφορετικό κόσμο, σαν να πρόκειται για μια χώρα η οποία συμμερίζεται τις αξίες μας σε σχέση με τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Είπατε ότι έγινε διαβούλευση με τα μέλη, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Δεν έχουμε να κάνουμε ε, με εταίρους που έχουν την ίδια αντίληψη με μας και την ίδια θέληση σε σχέση με αυτές τις βασικές αξίες. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, όπως είπε και ο κύριος Σέβιτς και ο Μάριο Νταβίδ. Δηλαδή ότι μιλάμε για, κοινωνία των, για κοινωνίες των πολιτών που ενισχύουν τις δημοκρατικές τους δομές και θα πρέπει να μάθουμε από την Τινησία. Δεν χρειάζεται να υποστηρίζουμε κυβερνήσεις που είναι δικτατορίες. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους λαούς. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει κάποιο ε, κάποιος συσχετισμός με τις ε, κυβερνήσεις, δηλαδή να έχουμε επαφή, αλλά να υποστηρίζουμε χρηματικά προγράμματα τα οποία επιτρέπουν την ελεύθερη έκφραση της γυναίκας στο σύστημα δικαιοσύνης, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με Ισλαμικές κοινωνίες, γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτό τον εκδημοκρατισμό μέσω των γυναικών και των νέων και να προβλέψουμε προγράμματα τα οποία θα αποτελέσουν σύνδεσμο της δικής τους ανάπτυξης με την ε, δική μας ολοένα και μεγαλύτερη ασφάλεια στις ανανεώσιμες κλιματικές αλλαγές, διατήρηση των υδάτων και ούτω καθεξής το θέμα της απασχόλησης των νέων είναι ύψης της σημασίας για μας αλλά και για εκείνους. Επίσης, ως προς τις συγκρούσεις, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι δεν, έχουμε θέση για τη Δυτική Σαχάρα. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό το θέμα. Είναι μια σημαντική σύραξη η οποία δυστυχώς δυσχεραίνει την, ε, την προσέγγιση Αλγερίας και Μαρόκου Κύριε Επίτροπε, ξέρετε πώς δίνονται χρήματα στη Δυτική Σαχάρα. Έχουμε, γιατί δεν είμαστε πιο απαιτητικοί από το Μαρόκο και το χρηματοδοτούμε. Και μπορείτε να σχολιάσετε την κατάσταση της νησία σε σχέση με τις γείτονες χώρες. Ναι, αυτό θα το δούμε και αργότερα. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο, έχετε να απαντήσετε σε πληθώρα ερωτήσεων. Ελπίζω να είσαστε σχετικά συνεκτικός. Thank you very much, Mr. Um, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω με σειρά γενικών σχολείων και στη συνέχεια θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Εκτιμώ ιδιαίτερο τη συζήτηση αυτή, γιατί δεν είναι απλώ ερωτήσει και απαντήσει. Η δική σα συμβολή και συνεισφορά πράγματι έχει μεγάλη αξία για μένα. Ε, τι θέλουμε. Θέλουμε η πολιτική γειτονία να γίνει ένα εργαλείο εταιρική σχέσης με τις κοινωνίες και όχι απλώς συνεργασία με αρχές ή εκπροσώπους αρχών. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, στο τέλος αυτής της διαδικασίας αναθεώρησης θέλουμε η πολιτική γειτονία να αντανακλά τα επιτεύγματα της Λισαβόνας. Α. Δεύτερον, να μας προσφέρει τη βάση ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφοροποίηση σε μεγαλύτερο βαθμό μεταξύ Νότου και Ανατολής. Και τρίτον, θα πρέπει να μας βοηθήσει να επιλύσουμε ένα ζήτημα. Να είμαστε δηλαδή συνεπείς αφενός, αλλά και ευέλικτοι από την άλλη, να μην πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο άκρο, αλλά να διαθέτουμε αρκετή ευελιξία και ευκαμψία ώστε να αντιδρούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Τρίτο σχόλιο. Η πολιτική γειτονία της Ευρώπης είναι μια εταιρική σχέση που εδράζεται στις αρχές της δημοκρατίας, ε, κράτους δικαίου, ε, χρηστής ε, διακυβέρνησης, σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, λέει ο μιλητή. Ταυτόχρονα ζητώ συγγνώμη που κάνω κακή χρήση των λέξεων. Η πολιτική γειτονία δεν είναι βραβείο Νόμπελ για μια καλή συμπεριφορά. Είναι ένα πρόγραμμα, είναι μια δέσμευση από δικής μας πλευράς να βοηθήσουμε τους εταίρους μας, τους γειτονές μας ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις. Και μάλιστα με τρόπο που τα ωφέλη θα φτάσουν στα κομμάτια εκείνα της κοινωνίας τα οποία το έχουν περισσότερη ανάγκη. Και παρακαλώ πολύ να γνωρίζετε ότι υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Οι αξίες μας, ο τρόπος διακυβέρνησής μας δεν είναι ο μοναδικός που προσελκύει το ενδιαφέρον των ε, γειτόνων μας. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Και το τέταρτο σχόλιο μου, γενικό μου σχόλιο κύριε Πρόεδρε, είναι ότι αυτό εγώ το θεωρώ ως έναρξη μιας επόμενης φάσης. Αυτή δηλαδή την ε, επικοινωνία ε, της διαδικασίας αναθεώρησης, μιας, μια ανταλλαγή απόψεων πάνω στην οποία θα συνεχίσουμε. Τώρα, έρχομαι σε πιο συγκεκριμένα θέματα. Ένωση για τη Μεσόγειο. Κύριε Σαλαφράγκα, Βάγκο, Μπίος κλπ. Συμμερίζομαι την ανησυχία σας. Και λυπούμε που βλέπω τον συνάδελφο, τον Γενικό Γραμματέα, να παρετείται σήμερα. Δεν μπόρεσα να μιλήσω μαζί του. Θα το πράξω το ταχύτερο δυνατό. Ήμουν εκεί στη Βαρκελόνη όταν εγγενιάσαμε τη γραμματεία και αμφότεροι μοιραζόμαστε αυτή τη φιλοδοξία, αυτό το όραμα της γραμματείας και αντιλαμβάνομαι το μέγεθος της απογοήτευσης που δοκίμασε. Αλλά η ουσία είναι ότι μία δεύτερη απόπειρα να διοργανωθεί μια διάσκεψη κορυφής απέτυχε. Χρειάζεται πολιτική καθοδήγηση, όθηση και ρωτάτε ποιοι χρηματοδοτούν τη γραμματεία, πόσες χώρες μέλη δεν είναι οι χώρες μέλη, είναι η Κομισιόν. Και δεν είναι ένα περιβάλλον το οποίο βοηθά τη γραμματεία να προχωρήσει και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο παρελθόν. Χρειάζεται πολιτικό momentum, χρειάζεται να υπάρξει μια νέα όθηση της συμπροεδρίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Δεν θεωρούμε τη Μέση Ανατολή ή τα θέματα της Μέσης Ανατολής ως προβλήματα που μας επιβάλλουν διαμεσολάβηση. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να κάνουμε μία ε, έξυπνη, να κάνουμε ένα έξυπνο συνδυασμό της ε, προσέγγισης μας με τις ε, κυβερνητικές επιλογές ώστε να απομονώσουμε τον ιό, να εστιάσουμε την προσοχή μας στην τομεακή συνεργασία όπου οι υπουργοί συνέρχονται και συμφωνούν πάνω σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Και έρχομαι στο ερώτημα του κυρίου Πάσκο. Ε, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Αλλά απλώς να πω ότι πήγα στην περιοχή, ε, επισκέφθηκα το Ισραήλ και τα κατεχόμενα και κάνω ό,τι μπορώ με τα κοινοτικά μέσα που διαθέτω για να προσφέρω στήριξη. Στον κύριο Μπάντου για το θέμα των χρημάτων. Η απάντηση είναι ναι και όχι. Εξαρτάται από τις φιλοδοξίες μας. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι δεν έχει να κάνει με περισσότερα χρήματα, αλλά έχει να κάνει με εξυπνότερη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων. Και αυτό συνδέεται και με την ευελιξία διότι ίσως δεν χρειάζομαι χρήματα στο πρόγραμμα Α, αλλά χρειάζομαι στο πρόγραμμα Β. Και δεύτερον, κοιτάξτε την Τινησία. Έχουμε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, για να τους βοηθήσουμε στις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό τομέα. Ε, το σχέδιο είναι για το 2013, αλλά πρέπει αυτό να γίνει στα τέλη του 11 αρχές 12, άρα χρειάζομαι μεγαλύτερη ευελιξία. Ταυτόχρονα έχει να κάνει με, τα, με αυτό που είπα, ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Οικονομική ολοκλήρωση. Αυτή η ε, βαθιά και ολοκληρωμένη συμφωνία που έχουμε. Ε, το έχω πει αρκετές φορές σε αυτή την Επιτροπή, ότι πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που επιτρέπει τους εταίρους να προσεγγίσουν τις νομοθεσίες τους και να προχωρήσουν σε πολύ βαθιές μεταρρυθμίσεις που κοστίζουν, που είναι δαπανηρές. Θέλουμε να είμαστε σοφαροί και θέλουμε να το πράξουν αυτό ώστε σταδιακά να γίνουν μέλη της εσωτερικής αγοράς. Και άρα πρέπει να αναζητήσουμε και να ανέβρουμε τρόπους για να τους στηρίξουμε και δεν θα πληρώσουμε γιατί το κάνουν για το δικό τους όφελος. Αλλά Ας πούμε ότι κάποιος έχει τις δυνατότητες αλλά είναι μόνος του. Και δεν έχει και το κίνητρο, ας πούμε, μιας μελλοντικής ένταξης σε εισαγωγικά. Άρα πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο. Κατανοώ λοιπόν την προσέγγιση σας σχετικά με τη χρηματοδότηση, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη και τις άλλες διαστάσεις, τις άλλες πτυχές. Συμφωνώ με το σχόλιο σας σχετικά με την άμεση δημοσιονομική στήριξη. Θέμα Ρωσίας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα πλέον να συνομιλήσουμε με τους γείτονες των γειτόνων μας. Δεν, η ομάδα στην οποία αναφερθήκατε δεν αποκαλείται πλέον φίλη της Ανατολικής Γειτονίας, αλλά είναι μια άτυπη ομάδα ε, συντονισμού και ενημέρωσης. Και στα τέλη ε, της, του περασμένου έτους η Ρωσία ζήτησε να είναι παρατηρητής, όχι πλήρες μέλος αυτής της άτυπης ομάδας. Αλλά το θέμα δεν συνδέεται μόνο με τη Ρωσία, αλλά και με άλλους σημαντικούς ε, εμπλεκόμενους σε αυτή την πολιτική. Προς τον κύριο Τένοκ. Ελπίζω ότι μετά από τέσσερα χρόνια θα είστε πιο αισιόδοξο από ό,τι σήμερα. Και ε, συμμερίζομαι κι εγώ την απογοήτευσή σας σε κάποιο βαθμό. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν σωστό να δει και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε αυτή η γειτονιά όλα αυτά τα χρόνια και ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Και πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν υπήρχε η ανατολική γειτονία και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για να προσελκύσουμε αυτούς τους εταίρους πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο ερώτημα του κυρίου Μποστινάρου σε σχέση με την Αλβανία, όπως γνωρίζετε, ένας απεσταλμένος της Κάθη Άστον βρίσκεται τώρα στην Αλβανία και είδαμε στην ουσία μία ε, συνέχιση του πολιτικού αδιεξόδου. Ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά στην ουσία δεν πρόκειται για εκλογές και εκλογική διαδικασία και ψηφοδέλτια. Το θέμα είναι πιο σοβαρό και ελπίζω οι ηγέτες και των δύο πλευρών να κατανοήσουν τις συνέπειες εάν συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία, δηλαδή αν ακολουθήσουν αυτή την πορεία. και ό,τι κάνουν τώρα ε, τίθεται κατά των συμφερόντων της Αλβανίας. Αποστήλαμε μία επιστολή λίγες μέρες πριν από την διαδήλωση αυτή. Δυστυχώς σκοτώθηκαν και αρκετοί άνθρωποι, κάτι το οποίο μας λυπεί ιδιαίτερα. Αποστήλαμε λοιπόν αυτή την επιστολή μιλώντας ε, για θέματα που απορρέουν από την έκθεση διεύρυνσης τονίζοντας ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των νέων εκλογών το Μάιο, των επικείμενων εκλογών και αναφέραμε ότι εάν δεν επιληθεί το θέμα αυτό, το πολιτικό καθαρά θέμα, δεν θα υπάρξουν ε, προπτικές διεύρυνσης, αλλά ακόμα χειρότερα είναι ότι θα υπάρξουν συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων. Και κινήθηκα και πέραν της παραδοσιακής μου στάσης και Μίλησα για το δείπνο πέρυσι τον Ιούνιο και είπα ότι βρισκόμαστε σε, μία, σε επαφή και με τις δύο οικογένειες και με τους δύο ηγέτες. Είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε και να επαναλάβουμε τη δέσμευσή μας εάν δεν μπορέσουν να αποφύγουν τα τελευταία προσκόμματα έτσι ώστε να φτάσουν σε μια πολιτική επίλυση του θέματος. Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι ότι ο Μύροσλαφ δέχεται, μάλλον την χάνει της υποστήριξης όλων των θεσμικών οργάνων και μίλησα με το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης με το Γενικό Γραμματεία του ΝΑΤΟ και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με κράτη ή διεθνείς οργανώσεις. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ενωμένοι σε σχέση με την αποστολή των μηνυμάτων αυτών. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι έχει περάσει ο χρόνος, αλλά νόμιζα ότι θεωρώ ότι πρέπει να επεκταθώ. Όσον αφορά τώρα την αναστολή της ε, σχέσης της ε, με τις χώρες ε, της πολιτικής γειτονίας προς Ανατολάς. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι η Λευκορωσία ακόμα δεν επωφελείται από το ότι μπορεί και αυτή να ενταχθεί στην πολιτική ανατολικής γειτονίας, αυτό είναι το τίμημα που καταβάλει η Λευκορωσία για το ότι δεν πράττει αρκετά τουλάχιστον όσον αφορά στο σεβασμό των αρχών αυτής της γειτονία. Ξέρετε ότι πριν από τις ε, εκλογές ε, εμείς ε, σκεπτόμασταν να τους προσφέρουμε ένα πολιτικό διμερές πλαίσιο για να υπάρχει κάποια εμπλοκή δική τους. Αυτό όμως δεν υπάρχει πια. Και την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσω τον Υπουργό Εξωτερικών για να συζητήσουμε και αυτό αλλά και άλλα θέματα. Και θέματα που είναι περιοριστικά αλλά και θέματα που αφορούν κυρίως στις ε, ανάγκες ε, των δημοκρατικών δυνάμεων και της ε, κοινωνίας. Αυτή η εταιρική σχέση μπορεί βεβαίως και να προσφέρει και ένα μικρό κομμάτι τεχνικής και οικονομικής βοήθειας. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό μπορεί να αποβεί τόσο χρήσιμο. Και επιπλέον <clears throat> πιστεύω ότι είναι σημαντικό το θέμα της Λευκορωσίας να μην αντιμετωπίζεται μόνο σε ένα θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Λευκορωσίας, αλλά σε ένα περιφερειακό θέμα πρέπει να μιλήσουμε και στους εταίρους μας, να μας πούν και εκείνοι πώς ακριβώς αισθάνονται μετά από αυτά που είδα στη τηλεόραση στις 19 Δεκεμβρίου. Και σιγά σιγά τελειώνω την παρέμβασή μου. Έχω μιλήσει επανειλημμένα για προστατευόμενες ε, σειράξεις. Σιγά σιγά ε, το να είναι κανείς ε, στο σημείο αυτό περισσότερο δραστήριος, αυτό βεβαίως ε, ε, καλύπτει τις, η συνθήκη της Λισαβόνας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <coughs> Eh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επέτρεψε να πούμε και πολλά άλλα, τα θέλαμε να το κάνουμε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Για να αποφύγουμε λοιπόν την ε, διασπάθηση χρόνου, ε, δεν θα πω τίποτα για το επόμενο θέμα και θα δώσω απευθείας ε, το λόγο σε εσά για να τοποθετηθείτε για το θέμα της τυνησίας και στο χρόνο που μας απομένει έχουμε μισή ώρα, μισή ώρα λέει ο πρόεδρος. που σημαίνει 10 λεπτά για σας και 20 λεπτά για μας. Κύριε Πρόεδρε. Ε, Όχι, δεν θα χωρίσω τη δήλωσή μου. Ε, δεν θα περικόψω, συγγνώμη, τη δήλωσή μου. Και θα την αναγνώσω, διότι μοιράστηκα κάποιες ε, ε, θέσεις ε, μαζί σας στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα και περιέλαβα και κάποια στοιχεία. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η Τινησία βρίσκεται σε μία καμπή της ιστορίας της σε έναν δρόμο προς την δημοκρατία. Μέσα σε λίγες μέρες ο πρόεδρος Μπενάλη εγκατέλειψε την ε, χώρα, το κόμμα του, το RCD διαλύεται, διαλύεται η Πολιτική Επιτροπή και μια μεταβατική κυβέρνηση διορίστηκε και περιλαμβάνει μέλη και της πρώην αντιπολίτευσης. Έχει ανακοινωθεί αμνηστία για όλους τους πολιτικούς κρατουμένους, έχει εξασφαλιστεί η ελευθερία του τύπου, και η απαγόρευση όλων των ομάδων υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αρθεί. Η μεταβατική κυβέρνηση διόρισε και μια επιτροπή με την εντολή να κάνει προτάσεις για πολιτικές μεταβολές οι οποίες πρέπει να γίνουν και δύο διαρευνητικές επιτροπές, μία για τη διαφθορά και μία για τις βιαιότητες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Αυτές είναι εξαιρετικές εξελίξεις και τις χαιρετίζουμε ολόψυχα. Ε, δημιουργούν ελπίδα για το λαό της Τινησίας που για μεγάλο χρονικό διάστημα έζησε χωρίς τη δυνατότητα να ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά του. Ωστόσο η Τινησία βρίσκεται απλώς στην αρχή της μετασχηματισμού της. Ε, ε, νέα μεταβατική κυβέρνηση θα χρειαστεί χρειαστεί τη δημόσια αποδοχή και οι αρχές της Τινησίας θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν τη δημόσια εμπιστοσύνη και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις στη μεταβατική περίοδο. Θα πρέπει να ξεκινήσει, να, επανεκκινήσει, να ξαναξεκινήσει η, η λειτουργία της οικονομίας και αυτό στο άμεσο μέλλον. Αυτή τη κρίσιμη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό του λαού της Τινησίας. Η Πατή Εκπρόσωπος και εγώ έχουμε ήδη προχωρήσει σε δηλώσεις, εκφράζουμε την υποστήριξή μας και τη βούλησή μας να έχουμε ανώτερα στελέχη της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στην Τινησία αυτή τη στιγμή που θα συναντηθούν με τις τρεις αυτές επιτροπές και με τους βασικούς παράγοντες περιλαμβανομένες της κοινωνίας των πολιτών και των ε, μελών της. Το επόμενο βήμα θα είναι μια επίσκεψη σε πολιτικό επίπεδο που ε, θα λάβει χώρα μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα συζητήσει το θέμα της Τινησίας ε, την επόμενη εβδομάδα και στην τελευταία ολομέλεια το σώμα αυτό συζήτησε το θέμα και ήμουν και εγώ παρόν. Επίση, αντιλαμβάνουμε ότι μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ταξιδέψει στην Τινησία πολύ σύντομα και το χαιρετίζω και αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι επιτροπέ του ω πολιτικά μέρη, ε, εταίροι σε διεθνέ επίπεδο έχουν σημαντικό ρόλο ώστε να συμβάλλουν στην θεσμική ενίσχυση των εταίρων τους της Ισία στο νέο περιβάλλον. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, τα αρχικά μέτρα που ανέλαβε η μεταβατική κυβέρνηση της Τινησίας είναι βήματα προς την ορθή κατεύθυνση και καλούμε τις αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τις νέες δεσμεύσεις ως προς τη διακυβέρνηση, το σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως επίσης και τη δέσμευση για κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη μεταβατική διαδικασία περιλαμβανομένης και της διοργάνωσης ελεύθερων, διαφανών και δημοκρατικών εκλογών το ταχύτερο δυνατό όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την πολιτική, νομική, τεχνική και υλική υποστήριξη που θα ζητήσει την Ισία για να προετοιμάσει και να οργανώσει τις εκλογές. Επίσης εξετάζουμε και άλλα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα υποστηρίξει την τη μετάβαση αυτή. Παραδείγματος χάρη, πάγωμα κεφαλαίων ατόμων που θα εντοπιστούν σε συνδυασμό με τις ε, νησιακές αρχές ε, προσαρμογή της χρηματοοικονομικής συνεργασίας μας στις νέες ανάγκες της χώρας και η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών της ε, Τινησίας. Θέλω να επιμείνω σε αυτό το σημείο, διότι είναι εμπειρία μας από οποιαδήποτε μεταβατική περίοδο, περιλαμβανομένης και της περιοχής από την οποία εγώ προέρχομαι στην Ευρώπη, ότι η κοινωνία των πολιτών χρειάζεται να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών ε, της Τινησίας από, Ευρωπαϊ... από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι απολύτως απαραίτητη, όπως είναι η πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία και τα προγράμματά μας για μη κρατικούς φορείς. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν μέσα από τα προγράμματα, την εταιρική σχέση, τα πολιτικά κόμματα, τα ιδρύματα και άλλους. Το βλέπω ως έναν από τους καλύτερους τρόπους να ενισχύσουμε το μέλλον της Τινησίας και να βοηθήσουμε τη σταθεροποίηση της δημοκρατίας το ταχύτερο δυνατό. Τώρα, ως προς την, ε, το καθεστώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις σε νέα βάση με ένα διάλογο με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και να συμφωνήσει σε ένα πρόγραμμα δράσης που θα είναι προσαρμοσμένο στη νέα κατάσταση. Είναι απόλυτα σαφές ότι το ενισχυμένο καθεστώς σημαίνει περισσότερη συνεργασία αλλά και πρόοδο σε θέματα όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταβάλει κάθε προσπάθεια υποστηρίζοντας την, την Ισία για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά της για να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που βρίσκονται στην ρίζα της δυσαρέσκειας έναντι του προηγούμενου καθεστώτος. Ανεργία και ιδιαίτερως η ανεργία που αφορά τους νέους και τους νέους πτυχιούχους. Η φτώχεια, η έλλειψη ανάπτυξης σε πολλές περιοχές της χώρας άμεση αντίδραση από πλευράς των νησιακών αρχών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ανοίξει η οικονομία, να διευκολυνθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, να αντιμετωπιστεί η διαφθορά, να ε, υπάρξουν ε, ε, να υπάρξει δανεισμός και να ενισχυθεί η οικονομία. Αυτά απαιτούν άμεσες μεταρρυθμίσεις. Κατά το παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την υποστήριξή της στους τομείς αυτούς και τώρα είμαστε έτοιμοι σε συνεργασία με τη δημοκρατική, ε, δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση να προχωρήσουμε. Η Τινησία είναι σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συμφέροντα ε, να υπάρχει μια ευημερούσα δημοκρατική Τινησία η οποία ε, θα Εποφεληθεί και αυτή και θα συμμετέχει σε αυτό το πλαίσιο που είναι οι κοινέ αξίες. Οι δικές μας οι οικονομίες είναι σταθερές. Ε, εμείς ε, λοιπόν ε, πρέπει να διαφυλάξουμε αυτά που επιτεύχθηκαν στο παρελθόν και να δημιουργήσουμε και νέες προποθέσει για το μέλλον. Είμαι λοιπόν δεσμευμένος ότι θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε μια δημοκρατική τιμησία η οποία θα μπορεί να είναι μοντέλο και ε, πηγή ελπίδας για τους λαούς ε, του ε, Μαγκρέπ και γενικότερα για ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Γρήγορα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση δύο λεπτά στον κύριο Σαλαφράνκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτά που είπε ο Επίτροπος είναι πολύ καθησυχαστικά και ε, βρίσκονται σε συμφωνία με αυτά που ελέγχθησαν και στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να παρακολουθήσει εξελίξεις, να στηρίξει τις ε, δημοκρατικές διαδικασίες, τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία, κυρίως στη δικαστική εξουσία για να λειτουργεί και αυτή αποτελεσματικά. Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να μάθουμε και νομίζω ότι έχει και σχέση με την πολιτική γειτονία. Να μάθουμε από τα λάθη που έχουμε κάνει. Διότι Μόνο έτσι θα επιτύχουμε τα ευκταία αποτελέσματα. Ε, έγινε λόγος για μια task force η οποία θα μπορούσε να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε αυτό καταλήξαμε στη συζήτηση ανάμεσα στις ε, πολιτικές ομάδες. Έτσι λοιπόν κύριε Επίτροπε θεωρώ ότι η δική σας στάση είναι πολύ καλή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύντομα νομίζω θα στείλει μια ad hoc επιτροπή και θεωρώ ότι οι δικές σας οι προσπάθειες και οι προσπάθειες της είπα ε, εκπροσώπου δείχνουν ότι δεν θα αποτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις φιλοδοξίες ελευθερίας, ε, της ε, την Αυτό είναι και προς δικό μας όφελος, το, προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαλαφράγκα. Μπιόρς για δύο λεπτά παρακαλώ. Η παρέμβασή σας μου φάνηκε τέλεια κύριε Επίτροπε. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Αυτή είναι η φωνή της Ευρώπης που θέλουμε να ακούμε σε αυτό το κοινοβούλιο. Δυστυχώς βέβαια η αντίληψη ε, των τινησίων ε, τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με το ρόλο της ε, Ευρώπης δεν ε, ήταν και ιδιαίτερα θετική. Πάντως πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να ισχυριστεί ότι έκανε κάτι. Βέβαια και η Επιτροπή. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η soft power της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και χρόνια είναι σε επαφή με τους δημοκράτες την ίσιους, με τους υπερασπιστές των, ε, της κοινωνίας των πολιτών και το, της ελευθερίας τύπου και των δημοκρατικών δικαιωμάτων στην Ισία. Έτσι λοιπόν, για να υπάρξει αυτή η μετάβαση, πρέπει να στηρίξουμε τους ετινήσιους. Παρότι λοιπόν σε αυτή την περίοδο της κρίσης υπήρξαν θετικές φωνές στην Ευρώπη, η την Ισία δεν ξέρω αν είναι κατά πόσον ρόλο της Ευρώπης έχει αποδώσει ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό που διακυβεύεται τώρα είναι η Μεσόγειος, οι σχέσεις ε, ανάμεσα στην Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο κατόπιν τούτου η τιμηθεία είναι καθοριστική σημασία. Και από εμά νομίζω θα εξαρτηθεί αν θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή σε επιτυχία, γιατί αυτό θα είναι καθοριστικό για την ευρύτερη περιοχή. Αν όμως από την άλλη τελικά η κατάσταση εξελιχθεί σε χάος, ε, θα επιδεινωθεί. Σάκε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε για την Τινησία, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αναφερθήκατε στην αβέβαιη κατάσταση και προσφέρατε βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όσο, παρά το γεγονό ότι είναι αβέβαιη η κατάσταση, είναι βέβαιο ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Κυρίω ε, ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι ελευθερίε των πολιτών. Και όσο και να διδαχθούμε, να διδαχθούμε ουσιαστικά από την, την Ισία. Χρειάστηκε να περάσουν 23 χρόνια δικτατορίας, τον οποία αποκαλούσαμε σύμμαχο, με πολύ σοβαρά φαινόμενα διαφθοράς και καταπίεσης, μάλιστα. Ε, και βέβαια προς το μέλλον της Τινησίας και οποιαδήποτε διαδικασία συμφιλίωσης, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη αλλά υπήρχαν διαφορές στις φωνές που ακούστηκαν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως μου έκανε εντύπωση η γαλλική κυβέρνηση Ελάχιστες ημέρες πριν από την πτώση της κυβέρνησης, η γαλλική κυβέρνηση εξέφρασε την υποστήριξή της προς ε, την ε, κυβέρνηση της Τινησίας. Πρέπει λοιπόν να διδαχθούμε από αυτά και καθώς εμείς ομιλούμε εδώ νεαροί ε, ξυλοκοπούνται στην Αίγυπτο, είναι μια γενιά η οποία ζητάει περισσότερες ελευθερίες, περισσότερα δικαιώματα, περισσότερες ελευθερίες και εμείς πρέπει να τους στηρίξουμε. Και ένας τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε και δεν το άκουσα από εσά και είναι σημαντικός, είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται αυτή η νέα γενιά παγκοσμίω και που ε, επιδεικνύει αλληλεγγύη μέσω του διαδικτύου ένα στον άλλον. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ε, ε, υπερβαίνουν δηλαδή τη λογοκρισία και χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία ε, και με αυτόν τον τρόπο ασκούν τα δικαιώματά τους μέσω των νέων τεχνολογιών. Πρέπει λοιπόν οι νέες τεχνολογίες να βρίσκονται στο στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντός μας, διότι και οι κυβερνήσεις είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να καταπιέζουν τους λαούς τους μέσα των τραφολόγιων. Ε, δύο λεπτά. Ε, κοιτάξτε, και εγώ ε, θέλω να απευθύνω έκκληση, γιατί έχω την εντύπωση ότι χάσαμε μία ευκαιρία. Αν περιμέναμε να δούμε ε, τι θα μας δώσει η καινούργια κυβέρνηση πριν να αν συνέβη κάτι πριν από 20 χρόνια θα είχαμε ένα σιδηρούν παραπέτασμα. Το θέμα είναι τι είδου ε, συνθήκες πρέπει να οριμάσουν για να στηρίξετε περισσότερο την κοινωνία των πολιτών, για να στείλετε σαφή μηνύματα στους νέους στην Τίνιδα και στην Αίγυπτο ότι είμαστε, σας στηρίζουμε. Νομίζω λοιπόν ότι στην Τινησία σήμερα θα μπορούσε να γίνουν πολλά περισσότερα. Η κυρία Άστον ε, θα μπορούσε από κοινού με τα Έθνη να στηρίξει τις ε, γυναίκες ως ε, σημαντικούς παράγοντες σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης θα μπορούσατε να βοηθήσετε να εξελιχθεί ο τύπος, να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία τύπου. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει, ε, ότι χρειαζόμαστε έναν ειδικό απεσταλμένο να πάει εκεί ε, και ε, να είναι το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν τα χρήματα να φτάνουν στο στόχο τους. Εμείς όσον αφορά τα 20 εκατομμύρια για το κράτος δικαίου τα καταργήσαμε, τα αρνηθήκαμε γιατί θα το μόνο για να απολυθούν κάποιοι δικαστές. Εμείς πρέπει λοιπόν να βλέπουμε ε, που ε, διοχετεύονται τα κονδύλια. Ε, πρέπει να αποδοθεί σημασία στην κοινωνία των πολιτών και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφερθήκατε στις επενδύσεις. δεν νομίζω ότι αρκεί να στηρίζει κανείς την εκλογική διαδικασία. Πρέπει να υπάρχει μια πιο βαθιά διαδικασία εγώ λοιπόν προτείνω να συστήσουμε μια ομάδα κρούσης ανάμεσα στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, για να υπάρξει αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο ε, χορηγούνται τα κονδύλια. Και ελπίζω ε, αυτή την ιδέα να την προάγετε. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με την κυρία Άουτολα για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, η δική μας υποπιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αποφασίσει ήδη να στείλει αποστολή στην, στην νησία όταν ακούσαμε το φθινόπωρο ότι το καθεστώς παίρνει πιο αυστηρά μέτρα. Και τώρα λοιπόν εμείς ε, ε, θα αποτελέσουμε ένα κομμάτι της ευρύτερη ε, αντιπροσωπείας που θα πάει στην νησία την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, τι είδους μέτρα πρέπει να ληφθούν για να στηριχθούν οι ε, νομοθετικές διαδικασίες. Κατανοώ ότι υπάρχουν πολλοί ε, κατασταλτικοί, καταπιστικοί νόμοι που πρέπει να τροποποιηθούν και μια χώρα ε, που πρέπει και θέλει να γίνει δημοκρατική χρειάζεται κάποιους θεσμού, όπως το διαμεσολαβητή παράδειγμα. Ίσως λοιπόν μπορούμε να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες σας για αυτό το θέμα και να μας συμβουλέψετε... Ε, για το πώς μπορούν να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Ε, μάλλον λάθος έκανα. Τον τελευταίο λόγο έχει ο κ. Χουντής. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να έχω τον τελευταίο λόγο, διότι όλα αυτά που είπε ο κύριος Φούλε ακούστηκαν τόσο ωραία που πίστεψε κανείς ότι είναι πραγματικότητα. Και επειδή ο κύριος Φούλε και προσωπικά η συνεργασία μας και η συνεργασία με την Επιτροπή και δεν αμφισβητώ τις προθέσεις μου, μου γεννήθηκε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Αν αυτή η συζήτηση γινόταν πριν ένα χρόνο, που είχαμε το καθεστώ Μπέναλι, τι θα μα έλεγε ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Ότι προθούμε αυτά, κάνουμε εκείνο κτλ. Το ερώτημα είναι, τόσα χρόνια υπήρχαν καταγγελίε για παραβιάσει τη δημοκρατία, για όλα, για διαφθορά κτλ. Και εμεί συνεχίζαμε μέσα στα πλαίσια τη καλή γειτονία και λέγαμε δεν τρέχει τίποτα. Τι εγγυάται, και δεν αναφέρομαι προσωπικά στον κύριο Φούλε, ότι αύριο δεν θα το έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Και λέω τι εγγυάται κανεί δεν μπορεί να σου δώσει υπόσχεση. Δεν έχω ακούσει όμω, λόγω, επιτρέψτε μου τη θρησκευτική έκφραση, μετανία, ότι εδώ κάναμε λάθο. Ότι κακώ αδιαφορήσαμε, κακώ ανοιχτήκαμε. Διότι κατά την άποψή μου από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δουλειές να γίνονται, οι πολυεθνικές να κερδίζουν και τα υπόλοιπα πηγαίνανε περίπατο. Ερώτηση πιο συγκεκριμένη. Πάμε για εκλογές. Έχει εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα των δυνάμεων που ήταν εκτός νόμου, των δυνάμεων της αριστεράς, αυτών που στράφηκαν και κυνηγήθηκαν από το καθεστώς Μπεναλή, Έχουμε εγγυήσεις ότι θα γίνουν τέτοιες ελεύθερες εκλογές. Τρίτη και ε, τελευταία ερώτηση. Ωραία, είπε ο κύριος Φούλε, να γίνουν ιδιωτικέ επενδύσεις. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι έχουμε εκτεταμένη φτώχεια, εκτεταμένη εξαθλίωση και δεν ξέρω πώς θα μπουν οι επενδυτές και οι επενδύσεις, δεν ξέρω πώς θα χρηματοδοτήσει και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν χρηματοδοτήσει ή βοηθήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις με το καθεστώς να γίνει εκμετάλλευση, ληστρική εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των άλλων ε, ε, ε, δυνατοτήτων που έχει η χώρα είναι φανερό ότι θα έχουμε νέες κοινωνικές εκρήξεις. Αν πάμε με την αίσθηση της αλληλεγγύης να λυθούν τα προβλήματα, ενδεχομένως να θεραπευθούν. Η τελευταία ερώτηση, επειδή δεν αναφέρθηκε. Ε, ποια είναι η εκτίμησή σας, κύριε Φούλε, δεν το πρόσεξα. Έχουμε το φαινόμενο της διάχυσης. Έχουμε την Ισία, Αίγυπτο και ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές. Μήπως αυτές τις αρχές πολιτικής γειτονίας σε ό,τι εξαρτάται την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα πάμε καλά, δεν έχουμε δώσει σωστά μηνύματα. Ευχαριστώ τελείως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Χουντή. Και βεβαίω ο τελικό λόγο, το λόγο θα δώσω στον κύριο Επίτροπο για να απαντήσει. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Uh, um, question. Σε σχέση με το τελευταίο ερώτημα, ως απάντηση σας ε, λέω ότι κάθε Άστον και εγώ ήμασταν αυτοί που δρομολογήσαμε την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Αυτή η πολιτική είναι μια διαδικασία. Διαδικασία όπου χρειάζεται να έχουμε και χρόνο να σκεφτούμε τα διδάγματα, τα όσα μαθαίνουμε στην πορεία. Και ως ένα βαθμό ε, έχουμε προβλέψει με την κάθε ότι χρειαζόμαστε αυτά τα νέα μέσα, μια νέα προσέγγιση έναντι αυτών των χωρών. Το ερώτημά σας, τι θα συνέβαινε πριν από ένα χρόνο. Μπορώ να σας πω ότι συνέβη πέρσι. με αυτό που συμφωνήθηκε με τις χώρες μέλη, δηλαδή λήφθη η απόφαση ότι χρειαζόμαστε μία διαδικασία η οποία θα καταλήξει στο νέο καθεστώς. Η πρώτη συνάντηση έγινε το Σεπτέμβριο πέρσι. Ήταν μία συνάντηση στο γραφείο μου με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Και συζητήσαμε το, την τροποποίηση του ποινικού κώδικα και ε, ποιοι συνεργάζονται και ποιοι δεν συνεργάζονται με την κοινωνία των πολιτών. Και αυτή η διαδικασία το Σεπτέμβριο πέρσι ξεκίνησε κάπως περίεργα. Εγώ στο μέσο αυτής της συνάντησης ζήτησα να μπω στην αίθουσα και να κάνω μία δήλωση, σύντομη δήλωση. Και στη δήλωση αυτή αναφέρθηκα στην αρχή που χρησιμοποιώ ξανά και ξανά ε, ενισχυμένο καθεστώς σημαίνει ενισχυμένες ε, ε, δεσμεύσεις και θέματα όπως το άρθρο 61 2 ε, και η κοινωνία των πολιτών δεν είναι συμβατά με το Βαντσέν. Και ε, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση της Τινησίας. Αυτά συνέβησαν πέρσι το Σεπτέμβριο. Δεν έχουμε απλώ τα ανώτερα στελέχη τη υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και ούτε ζήτησα και την άδεια από την κάθη για να κάνω αυτή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, αλλά θα το κάνω ως διευθύνων σύμβουλος αν θέλετε, managing director. Χωρίς μικρόφωνο το σχόλιο. Είναι Managing Director, Διευθύνων Σύμβουλος, που σημαίνει ότι είναι υπεύθυνος για την πολιτική στις χώρες αυτές. Σε αυτό τον υψηλό και σημαντικό ρόλο είναι ο καλύτερα εξοπλισμένος, αν θέλετε, για να ε, αποτιμήσει την κατάσταση επιτόπου. Είπα ότι θα μιλήσει με τους εκπροσώπους των τριών επιτροπών, περιλαμβανομένης και αυτής, η οποία είναι επιφορτισμένη με την προετοιμασία των εκλογών και θα προτείνει τις διάφορες αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ε, αλλαγές, δύσκολες αλλαγές στην νομοθεσία. Ήδη έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να αποστείλουμε έναν εμπειρογνώμονα που θα βοηθήσει στην τροποποίηση της νομοθεσίας. Και όταν επιστρέψει, ασφαλώς θα έχουμε ενδεχομένως την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και τότε θα, ίσως θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Στη, με τη συγκεκριμένη δική σας υποεπιτροπή, αλλά και με το Κοινοβούλιο γενικότερα και ασφαλώς μπορεί να βοηθήσει το Κοινοβούλιο. Και ασφαλώς θα περάσω το μήνυμα σχετικά με την ομάδα δράσης, την Task Force. Το αν θα υπάρξει η ομάδα δράσης ή όχι είναι ένα θέμα, αλλά πρέπει να πω ότι αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία που συζητούμε την Τινησία, η δεύτερη φορά και εικάζω ότι σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον και ελπίζω ότι αυτή η στενή επικοινωνία μεταξύ μας και, με, και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Κομισιόν και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σωστά προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, λέει ο Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφου. Οι παρεμβάσει ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη ε, συνάντησή μα με θετικά ε, θετικές εικόνες. Ελπίζουμε η συνεργασία να είναι εποφελής και ε, νομίζω ότι πράγματι όλα αυτά που γίνονται τα εκτιμούμε ιδιαίτερα. Όπως ξέρετε λοιπόν, προβλέπετε αυτή η ad hoc αντιπροσωπεία, το είπατε κι εσείς, η οποία θα φύγει μετά τη συζήτηση στην Ολομέλεια και ελπίζω εκεί να μπορέσετε κι εσείς να διαδραματίσετε το ρόλο που θα θέλατε, όπως είπατε σήμερα. Έγινε ήδη μια συζήτηση σε μια συνάντηση που είχαμε. Εμείς προσφέραμε την βοήθειά μας και θεωρώ ότι θα μπορούσε πράγματι να υπάρχει και μια επιτροπή ε, παρακολούθησης ε, των εκλογών γιατί από ό,τι φαίνεται σε 60 ημέρες ε, θα υπάρξουν εκλογές στη χώρα αυτή και ευχόμεθα οι εκλογές να είναι δημοκρατικές. Σας ευχαριστώ όλους σας. Να σας κάνω και μια τελευταία ανακοίνωση όσον αφορά την κατάθεση των τροπολογιών για την έκθεση ε, σχετικά με την Μεσόγειο μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου στις 12. Αυτή είναι η καταλεκτική ημερομηνία. Ε, και μόνο στα αγγλικά γιατί δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και γεια σας.